Αγαπητοί συναδελφοί, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ήδη περιμέναμε 15 λεπτά, 10 λεπτά. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στη συνεδρίαση αυτή. Να σας πω ότι ε, ω συνήθως μεταδίδεται από το διαδίκτυο συνεδρίαση αυτή. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι αν ε, η συζήτηση με τον ε, Υφυπουργό κύριο Μαυρογιάννη τελειώσει νωρίτερα, μπορούμε από σήμερα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τις ε, οδηγίες και τους κανονισμούς που έχουμε στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Δεν έχω λάβει καμία πρόταση για τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης. Έκανα μόνο αυτό το μικρό σχόλιο από τη δική μου την πλευρά. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι υπάρχει ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης και ενδεχομένως να πρέπει να κάνουμε κάποιες ε, προσαρμογές εφόσον ε, χρειαστεί. Δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη ανακοινώσει της Προέδρου. Δεν έχω να κάνω κάποια ανακοίνωση. Περνάμε λοιπόν στο τρίτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Δεύτερη ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα της Κύπρου, ο οποίος είναι Προεδρεύων του Συμβουλίου, με τον κύριο Ανδρέα Γιάννη, ο οποίος θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες όσον αφορά το, το μελλοντικό έργο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, το έργο το οποίο γίνεται για τα νομοθετήματα που μας αφορούν και ένα γενικότερο απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας. Έχετε το λόγο κύριε Υφυπουργέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Τελευταία φορά που παίρνω το λόγο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, θα ήθελα λοιπόν να σας πω Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο κομπλιμέντο, αλλά το λέω ειλικρινά ότι ένα από τα πράγματα τα οποία θα μου λείψουν είναι πολύ ιδιαίτερη και παραγωγική επικοδομητική σχέση που είχα μαζί σας με τη δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, και από τις δύο πλευρές θα κρατήσουμε μια πάρα πολύ θετική ανάμνηση της ε, πολύ καλής αυτής συνεργασίας που είχαμε τους τελευταίους έξι μήνες. Ξέρετε ότι κάθε φορά στα πλαίσια μιας Προεδρίας Χαίρεται κανείς πάρα πολύ όταν στο τέλος της Προεδρίας, μάλλον χαίρεται κανείς που αναλαμβάνει την Προεδρία, αλλά χαίρεται ακόμα περισσότερο όταν ολοκληρώνεται η Προεδρία αυτή. Έχουμε μπει λοιπόν ήδη σε νεορταστικό, χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Πρέπει όμως να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων, να έχω αυτή την ανταλλαγή απόψεων μαζί σας, προτού ολοκληρωθεί η Κυπριακή ε, Προεδρία. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ, στην αίθουσα αυτή για δεύτερη φορά και θα ήθελα πολύ γρήγορα να κάνω ένα σύντομο απολογισμό των επιτευγμάτων της Κυπριακής Προεδρίας στο τελευταίο εξάμεινο. Θα ήθελα καταρχά να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα, να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι επιτροπέ του για την ενεργή συμμετοχή, καθώ επίση και για τη συμβολή του, ιδίω όσον αφορά τι συζητήσει για τα ζητήματα τα οποία βρίσκονται αυτή, αυτή τη στιγμή εξέλιξη προκειμένου να δημιουργηθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα διέπει τι πρωτοβουλίε και τι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020. Μια πολύ αξιοσημείωτη εργασία έχει γίνει από τι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ και ιδίω από τη δική σα την επιτροπή, η οποία πολύ σημαντικά συμβάλλει στην επιτυχή έκβαση της εργασίας κάθε Προεδρίας του Συμβουλίου στα ζητήματα εκείνα τα οποία πετούν απόφαση. Όταν έκανα την πρώτη παρουσίασή μου τον Ιούλιο, παρουσιάζοντα το πρόγραμμα τη Κυπριακή Προεδρία, αναφέρθηκα στην εργασία την οποία γίνεται για να δημιουργήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη για τι επόμενε γενιέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στο μέλλον μια Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγαλύτερη σημασία για του πολίτε και τον κόσμο, που να μπορεί να συμβάλλει πιο αποτελεσματικά στην αηφόρο ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασία και να δημιουργεί υψηλότερα ποσοστά αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή καταπολεμώντας την αυξανόμενη ανεργία των νέων. Όλα αυτά αποτέλεσαν για μας βασικούς στόχους και βασικές προτεραιότητες. Όσον αφορά τώρα τις ιδιαίτερες προτεραιότητες που πρέπει να μας απασχολήσουν κατά δεύτερο εμείς του 2012, πρέπει να σας πω ότι η Κυπριακή Προεδρία έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχή διαχείριση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου με στόχο να πετύχουμε έναν από τους βασικούς στόχους της Προεδρίας, δηλαδή την πρόθεση μιας πιο αποτελεσματικής και βιώσιμης Ευρώπης. Μετά την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενδιάμεση έκθεση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, η Κυπριακή Προεδρία τον Οκτώβριο 19 Οκτωβρίου πρότεινε ένα δεύτερο διαπραγματευτικό πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνονταν για πρώτη φορά αριθμητικά στοιχεία και γινόταν μια εξισορροπημένη πρόταση η οποία αντικατόπτριζε τα θέση των κρατών μελών καθώς επίσης και συμβασμούς που είχαν ευρεθεί μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κρατών μελών και λάβαμε βέβαια υπόψη και τη σημαντική συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις αρχές Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέλαβε τις επραγματεύσεις για το πολιτές νομοσνομικό πλαίσιο με όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη πρόταση λοιπόν που έκανε ο πρόεδρος Ροπόη είχε ως στόχο να πετύχει μια ισορροπία με διαφορετική όμως προσέγγιση. Ενώ στη δεύτερη του πρόταση, την οποία παρουσίασε κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ήρθε πιο κοντά στην πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας. Θεωρούμε ότι κατά τη διάρκεια της ε, συνεδρίασης αυτής βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Οι αρχηγοί κρατός και κυβερνήσεων είπαν ότι θέλουν στις αρχές του 2013 να πετύχουν μία συμφωνία. Παράλληλα, η Κυπριακή Προεδρία θέλησε να σημειωθεί πρόοδο σε κάποιε κοινέ πολιτικέ και κοινά προγράμματα στα πλαίσια του διεθνού νομισμα... του, διεθνούς, του πολιτισμού με δημοσιονομικού πλαισίου, ιδίως όσον αφορά τις βασικές προτεραιότητες για την στρατηγική Ευρώπη 2020. Αρχίσαμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε πιο έντονα ακόμα με τα κράτη-μέλη και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε μία συμφωνία για τις νομοθετικές προτάσεις και προκειμένου η τομεακή νομοθεσία να εγκριθεί εγκαίρως. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να επικεντρωθούμε στην πολιτική συνοχή. Όταν συνεδριάσαμε τον Ιούλιο, σας είπα πόσο σημαντική ήταν η πολιτική αυτή για την Προεδρία μας και είχαμε πει τότε ότι δεσμευόμασταν προκειμένου να διευκολύνουμε μια έγκαιρη συμφωνία για το νομοθετικό αυτό πακέτο για τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Επαναλάβαμε τη δέσμευση αυτή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας που έλαβε χώρα στη Λευκοσία το Σεπτέμβριο, στα πλαίσια της επίσκεψης της αποστολής της Επιτροπής σας στην Κύπρο. Συνεχίζοντας με εμείς μετά την Δανέζικη Προεδρία, ξεκινήσαμε ως Κυπριακή Προεδρία με ένα πολύ έντονο πρόγραμμα στα πλαίσια του Συμβουλίου, έχοντας ως στόχο να ολοκληρώσουμε όλα τα εκκρεμή ζητήματα τα νομοθετικά μέχρι το τέλος του 2012 με την εξαίρεση των χρηματοπιστωτικών ζητημάτων που εξαρτώνται από την έκβαση των πραγματεύσεων για το πολιτές νομοσυνομικό πλαίσιο. Τα πρώτα αποτελέσματα τα είδαμε τον Οκτώβριο με κάποια συμβαστικά κείμενα για 7 θεματικά νομοθετήματα τα οποία είχαν συμφωνηθεί σε μια πρώτη φάση από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στα ζητήματα της εδαφικής ανάπτυξης, της ε, Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πληροφόρηση, την επικοινωνία, με συγκεκριμένου δείκτε και με χρηματοπιστωτικά ζητήματα τα οποία βρίσκονται εκτό πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Αναφερθήκαμε, για παράδειγμα, στη διαφοροποίηση τη ε, χρηματοδότηση και στην αρχή τη προστατικότητα. Στη συνέχεια, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Νοεμβρίου προχωρήσαμε περισσότερο με δύο ακόμα διαπραγματευτικά πλαίσια, με την ε, χρηματοπιστωτική διαχείριση καθώ επίση και με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο το οποίο συζητήθηκε ως παράρτημα του κανονισμού για τις κοινέ διατάξεις. Με μια τροποποιημένη πρόταση το Σεπτέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενσωμάτωσε μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου στον κανονισμό κοινών διατάξεων, ενώ η Κυπριακή Προεδρία μέσω των συμβαστικών κειμένων, τον οποίο πρότεινε, κατάφερε να ενσωματώσει το κοινό στρατηγικό πλαίσιο στο σύνολό του, στα πλαίσια του ε, παραρτήματος του κανονισμού κοινών διατάξεων, δίνοντας ένα πολύ συγκεκριμένο στρατηγικό προσανατολισμό στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο, μετά από αίτημα των κρατών μελών. Ανάλογη προσέγγιση έκανε και η δική σας Επιτροπή τον Ιούλιο. Μετά από τη συμφωνία που ε, επετεύχθη για τα δύο ε, επιπλέον νομοθετικά πλαίσια τον Νοέμβριο, ξεκινήσαμε τριμερείς διαλόγους όσον αφορά τους ε, κανονισμούς κοινών διατάξεων και από τον Εύρο και μετά όσον αφορά τον κανονισμό για τα ταμεία, για τα επιμέρους ταμεία, βλέποντας όλα τα θεσμικά όργανα τελικά ότι χρειαζόμασταν ε, συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις εγκαίρως, προκειμένου να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε εγκαίρως τα νέα προγράμματα ε, πολιτικής συνοχής στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειές τους. Σε σχέση με τους άτυπους αυτής τρισμερούς διαλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για το πνεύμα συνεργασίας το οποίο καταδείξανε τα θεσμικά μας όργανα, καθώς επίσης και την ταχύτητα με την οποία οι διαπραγματεύσεις αυτές ε, ολοκληρώθηκαν. Η Κυπριακή Προεδρία υπέβαλε στο Συμβούλιο σε πάρα πολλές συζητήσεις που είχαμε πέντε ε, συγκεκριμένες προτάσεις με τις οποίες ασχολήθηκαν οι πέντε επιμέρους διαπραγματευτικές ομάδες στα πλαίσια των συζητήσεων που έλαβαν χώρα για τον καονισμό κοινών διατάξεων και τον καονισμό για τα ταμεία. Συγκεκριμένα μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, 9 τριμερείς διάλογοι είχαν ξεκινήσει για τον καονισμό κοινών διατάξεων, 3 τριμερείς διάλογοι για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 3 τριμερείς διάλογοι για την ε, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, ένας τριμερείς διάλογος για τον κανονισμό του Ταμείου Συνοχής, καθώς επίσης και 6 τριμερεί διάλογοι για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τον στρατηγικό προγραμματισμό το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να δοθεί μια ασφάλεια δικαίου στα κράτη-μέλη για την προετοιμασία και την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Πιστεύω ότι ήδη έχουμε καλύψει ένα πολύ σημαντικό μέρο τη εργασία που πρέπει να κάνουμε και οι συνομοθέτε θα καταλήξουν, πιστεύω, πάρα πολύ γρήγορα σε μια συμφωνία όπω φάνηκε και στον τριμερή διάλογο τη προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα λοιπόν για όλη αυτή την πρόοδο να ευχαριστήσω του Ευρωβουλευτέ και ιδίω όσου συμμετείχαν στι ομάδε διαπραγμάτευση. Η Κυπριακή Προεδρία κατέβαλε πολύ σημαντικές προσπάθειες μέσα από την προετοιμασία κειμένων μέσω έντονων συζητήσεων προκειμένου να καταλήξουμε στον λεγόμενο πίνακα τεσσάρων στυλών. Τα κράτη-μέλη, τα οποία συμμετείχαν στις ομάδες εργασίες κατέδειξαν στην Προεδρία ότι ήταν σε θέση να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς όσον αφορά το στρατηγικό προγραμματισμό για το κανονισμό κοινών διατάξεων και για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχε μια κοινή βάση συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα θεσμικά όργανα. Πιστεύουμε ότι αυτή την εβδομάδα, τη 19η Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, η Κορεπέρ θα δώσει στην Προεδρία την απαραίτητη εντολή προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια σε μια προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στα δύο θεσμικά όργανα. Η Προεδρία στη συνέχεια θα υποβάλει στην Κορεπέρ μια έκθεση προόδου όσον αφορά του τρεμερού αυτού διαλόγου που ξεκίνησαν υπό την ε, Κυπριακή Προεδρία. Θα ήθελα επίση να σα πληροφορήσω ότι σε σχέση με τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι διαπραγματεύσει με την Επιτροπή Απασχόληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν προχωρήσει πολύ, σε τέτοιο μάλιστα σημείο που μπορεί να επιτευχθεί μια προκαταρκτική συμφωνία πολύ σύντομα ανάμεσα στα δύο θεσμικά όργανα. Θα ήθελα τώρα να επαναλάβω τη σημασία των εξελίξεων αυτών που θα δώσουν στα κράτη-μέλη και στι περιφέρειες μια ασφάλεια δικαίου, προκειμένου να καταφέρουν να προχωρήσουν ναι, περισσότερο τις προετοιμασίες τους για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Επίσης πιστεύουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο αποστέλουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς τον Ευρωπαίο πολίτη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να βοηθήσει τις περιφέρειες να κάνουν επενδύσεις και κατά αυτόν τον τρόπο να βγουν από την κρίση, λαμβάνοντας υπόψη τον εργό ρόλο όλων των εμπλεκομένων εταίρων. Τέλος, όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τα νομοθετήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική συνοχή και τη σχετική εργασία που έκανε η Κυπριακή Προεδρία, θα ήθελα να αφαιρθώ λίγο στι συνεδριάσει αυτέ που οργανώθηκαν στην Κύπρο, αρχή γενομένη από το Σεπτέμβριο, όπου είχαμε συνεδριάσει των ομάδων εργασία στα πλαίσια τη διακυβερνητική συνεργασία για ζητήματα εδαφική και αστική συνεργασία. Οι συναντήσει αυτέ ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο με την άτυπη συνεδρία των Υπουργών Αρμοδίων για την Πολιτική Συνοχή. Η Κυπριακή Προεδρία κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες προκειμένου να προχωρήσουμε περισσότερο με τα ζητήματα εδαφικής συνοχής. Στόχος της Προεδρίας ήταν να συμβάλλει πολύ στον τομέα αυτό, συνεχίζοντας την πολύ καλή διακυβερνητική συνεργασία η οποία υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οργανώθηκαν πάρα πολλέ συνεδριάσει σε επίπεδο τεχνικό αλλά και σε επίπεδο γενικών διευθυντών. Όλα αυτά καταδεικνύουν την πολύ μεγάλη σημασία που δίνει η Κυπριακή Προεδρία στην εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής. Διοργανώθηκαν μάλιστα συναντήσεις γενικών διευθυντών τόσο για ζητήματα εδαφικής συνοχής όσο και για ζητήματα πολιτικής συνοχής και προτιμάσαμε κατά αυτόν τον τρόπο την άτυπη υπουργική συνεδρίαση του Νοεμβρίου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες προκειμένου να ενσωματωθεί η εδαφική συνοχή όλο και περισσότερο στις εθνικές και κοινοτικέ πολιτικές και θα πρέπει να διατηρήσουμε επίσης και τη δυναμική της διακυβερνητικής αυτής συνεργασίας. Αυτά, αν θέλετε, είναι και τα δύο βασικά συμπεράσματα των όλων συζητήσεων που έγιναν. Όσον αφορά τώρα την άτυπη συνεδρίαση υπουργών του Νοεμβρίου, θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως την κυρία Χούμπνερ για την παρουσία της στη συνεδρίαση αυτή και για την πολύτιμη συμβολή της συζητήσεις που έλαβαν χώρα και οι οποίες επικεντρώθηκαν στην αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης της αναθωρημένης πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020. Ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας που έγινε για τη διακυβέρνηση της πολιτικής συνοχής και κοινοτικό επίπεδο ήταν η προστιθέμενη αξία του να έχουμε ένα συστηματικό πολιτικό διάλογο για την πολιτική συνοχής και για τις συμπεράσματα της πολιτικής αυτής σε επίπεδο Συμβουλίου. Κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι μπορεί να βελτιωθεί η σχετική διακυβέρνηση και να επεκταθεί περισσότερο η αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής. Η δυνατότητα διασύνδεσης της συζήτησης αυτής με την νέα κοινοτική οικονομική διακυβέρνηση και με το ευρωπαϊκό εξάμεινο εξετάστηκε. Η βασική έκβαση των συζητήσεων αυτών και της άτυπης υπουργικής ε, συνάντησης συνοψίζονται στα συμπεράσματα της Προεδρίας, τα οποία συμπεριλήφθησαν στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων που έλαβε χώρα στις 20 Νοεμβρίου. Τέλος, η Κυπριακή Προεδρία ζήτησε μια γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή όσον αφορά την ε, σημασία της δημιουργίας μιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής για την Μεσόγειο. Η θετική γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ υπερψηφίστηκε στην ε, Ολομέλεια της ΕΟΚΕ τον Νοέμβριο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Έχοντας κάνει έναν απολογισμό της εργασίας της Κυπριακή Προεδρία του τελευταίου έξι μήνε, μπορώ να πω ότι από κοινού έχουμε συμβάλει προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδο στον τομέα αυτό. Πιστεύω ότι αυτή την αξιολόγηση κάνετε κι εσείς για την κοινή μας συνεργασία και όπως είπα στην αρχή της παρεμβασής μου, θεωρούμε ότι ε, η πολύ επικοδομητική συνεργασία της δικής σας Επιτροπής προς την Προεδρία έχει συμβάλει πάρα πολύ σημαντικά στην πρόοδο αυτή. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρετε να συνεχίσετε και με την Ιρλανδική Προεδρία στο ίδιο επικοδομητικό πνεύμα. Από ό,τι έχω καταλάβει και η Ιρλανδική Προεδρία θέλει και αυτή να ολοκληρώσει τα νομοθετικά αυτά ζητήματα το στομότερο δυνατό. Ελπίζω θα καταφέρουμε να πετύχουμε μια έγκαιρη συμφωνία για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και ότι θα καταφέρουμε πολύ γρήγορα να εγκρίνουμε και το νομοθετικό πακέτο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πολιτική Συνοχή. Κυρία Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Thank ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Συνάδελφοι, να σας πω επίσης πως ε, βρίσκεται εδώ πέρα και ο Αντώνης Κωνσταντινίδης. Όσοι διαπραγματευτήκατε μαζί του στον διμερή διάλογο τον γνωρίζετε. Αντιλαμβάνομαι πως ε, ο κύριος Υπουργός ε, θα δεχτεί και ερωτήσεις αν υπάρχουν. Ο Λαμπέρ Φανίστελ Ρόι βλέπω είναι ήδη έτοιμος. Σύντομα, γιατί και άλλοι συνάδελφοι θα παρέμβουν. Δεν θα είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα όσο την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, από που βγήκατε αλόβητος. Τώρα, για την συνεργασία και το πνεύμα της συνεργασίας το οποίο φέρατε. Για να είμαι ειλικρινής, ε, είναι κάτι ε, το οποίο μαθαίνουμε και εμείς, οι βουλευτές, μαζί με το Συμβούλιο κάναμε τις εσωτερικές μας διαπραγματεύσεις, ε, την εντολή, την ψηφοφορία και μετά μάθαμε πως η άλλη πλευρά, το Συμβούλιο, είχε μία ανάλογη διαδικασία. Αλλά βεβαίως ε, ανέμπαινε το Συμβούλιο πως θα πιστεί πιο εύκολα το Κοινοβούλιο, αλλά αυτό δεν συνέβη. Και Βεβαίω ε, τα εξηγούσαμε, εξηγούσαμε ο ένας ε, τις θέσεις του στον άλλον και αυτό ήταν αναγκαίο. Γιατί πραγματικά μιλάμε για τις βασικές επενδυτικέ πολιτικές για την ε, επόμενη δεκαετία και χρήστηκαμε κάποιο χρόνο και μετά από λίγο καταλήξαμε σε μια φάση συμφωνίας ε, γνωρίζοντας πως ε, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο έχουν τις ίδιες ε, νομοθετικές αρμοδιότητες. Αυτό πρέπει να το λέμε καμία φορά. Και εντωμεταξύ συμφωνώ σημειώθηκε αυτή η πρόοδος και νομίζω πως φέτος θα μπορέσουμε να έχουμε μια μερική συμφωνία και για το στρατηγικό σχεδιασμό και την θεματική συγκέντρωση και το στρατηγικό πλαίσιο. Οπότε αυτό, αυτά τα οποία υποσχεθήκατε έγιναν και επίση για τους άλλους ε, κανονισμούς, για τα συγκεκριμένα ταμεία, είχαμε μια γρήγορη αρχή τους τελευταίους μήνες και νομίζω, όταν τα κοιτάμε αυτά, εξακολουθεί να ισχύει πως είμαστε πόροι, αν δείτε τον τομέα της γεωργίας, της αλίας, δεν ψήφισαν καν. Οπότε μαζί με το Κοινωνικό Ταμείο και την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης είμαστε πρωτοπόροι σε αυτή τη συζήτηση. Και δεν είναι άσχημο το ότι ε, βλέπουμε τις νέες μας αρμοδιότητες και βλέπουμε πώς πάνε τα πράγματα. Οπότε κάνετε καλά τη δουλειά σας, θα έλεγα εγώ. Θα ήθελα τώρα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τη γενική κατάσταση. Βεβαίω είπατε πως είμαστε κοντά σε μια συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά εξακολουθεί να έχουμε μια ε, περικοπές άνευ προηγουμένου στην πολιτική συνοχής. Οπότε καλό είναι το ίσως το ότι δεν έχουμε συμφωνία τώρα. Καθώς ε, δεν νομίζω πως μπορούμε να, να επιστρέψουμε, να, να από τώρα μέχρι το Ιαρινό Συμβούλιο. Όσες χώρες ε, θέλουν να πιστοχωρήσουν ε, μπορούν να αναπερικόψουν ε, τα δικά τους κονδύλια στο μέλλον. Αυτό, αυτό ήθελα να πω. είναι κρίμα, αλλά ελπίζω να μην έχουμε άλλες περικοπές σε αυτό το τομέα. Και το δεύτερον, Ξεκολουθούμε ακόμα να διαπραγματευόμαστε με βάση τις εντολές μας, αλλά το Συμβούλιο έχει τόσες ε, ευθύνες ε, που έχουν μπει σε αυτό το διαπραγματευτικό κουτί του Κούδεπου, ε, έτσι ώστε δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί τα σημαντικά μπαίνουν βεβαίως στο διαπραγματευτικό κουτί και πρέπει να τα διαπραγματευτείτε με την Επιτροπή μας και αυτό ακόμα δεν έχει συμβεί. Θα τελειώσω λέγοντας πως κάνατε εξαιρετική δουλειά μαζί με τους βοηθούς. Τους βοηθούς σας στις ε, διαπραγματεύσεις και δεν είναι πάρα πολύ αργά ε, για να καταλήξουμε σε σωστούς ε, καλούς συμβασμούς για τα κεφάλαια που δεν έχουμε ολοκληρώσει και βεβαίως Αναμένω πως ε, στον αφορά την πολιτική συνοχής ε, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα του χρόνου με τους Ιρλανδούς και μετά θα πάμε στην Ολομέλεια. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ. Κωνσταντσε Ευχαριστώ Ντανούτα. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα όσα είπε ο Λάμπερτ. Συμφωνώ με όλα. Δύο πράγματα θα ήθελα να τονίσω. Πρώτον, να ευχαριστήσω όλους όσους ε, συνσέφεραν έτσι ώστε να καταλήξουμε κάπου με το πρώτο πακέτο του στρατηγικού προγραμματισμού και βεβαίως ε, και την διαπραγματευτική ομάδα γιατί ξεκαθαρίσαμε πως ε, ήμασταν τελείως ε, διάφανοι σε όλη τη διαπραγματευτική διαδικασία. Δεν πήγαμε κάπου, ας μόνοι μας εγώ και ο Λάμπερτ. Ήταν μια απόφαση όλων γιατί για εμάς ήταν ξεκάθαρο όταν ξεκινήσαμε με τον τριμερή διάλογο πως οι θέσεις μας ε, που είχαμε ε, ψηφίσει ήταν μια θέση διαπραγματευτική. Οπότε δεν θα είχαμε ως αποτέλεσμα 100% την εντολή μας. Ε, έπρεπε να βρεθούν κάποιοι συμβιβασμοί και ήταν κάτι το οποίο κάναμε βεβαίω δημοσίως. Και επίσης Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την γραμματεία, τους συνεργάτες, ε, τους πολιτικούς συμβούλους, ε, όλους όσους βοήθησαν σε αυτό. Και μάλιστα εξεπλάγει κάπως για το ότι παρά το ότι ξεκαθαρίσαμε πως είμαστε στην διαδικασία της ε, συναπόφασης, είχα την εντύπωση πως ε, τα κράτη-μέλη αλλά και η Κομισιόν καμιά φορά ε, εκπλήσονταν αυτό ότι ε, εμείς παίρναμε στα σοβαρά αυτή την διαπραγμάτευση. Εγώ ήμουν σε εννέα γύρους διαπραγματεύσεων και βέβαια η διαδικασία αυτή θα είχαν πάει πάρα πολύ γρήγορα εάν όλοι το έβλεπαν ως μια πραγματική διαπραγμάτευση και δεν έλεγαν ότι θα αποφασίσουν τα κράτη-μέλη και μετά α, θα το δεχτεί το Κοινοβούλιο. Άλλαξαν λοιπόν τα πράγματα, ίσως να είναι απλούστερα την επόμενη φορά, γιατί τα κράτη-μέλη ξέρουν πώς πρέπει να κινηθούν, αλλά τελικά τα καταφέραμε μαζί και είναι ενδιαφέρουσα η εμπειρία, το πώς δηλαδή θα ε, μπει μια δυναμική στη διαδικασία. Αυτό το οποίο θα ήθελα να επαναλάβω εδώ πέρα και ευχαριστώ και την Προεδρία. Ε, ναι. Το εξή. Ε, στο κέντρο πρέπει να είναι και για μας και για την Κομισιόν και για τα κράτη-μέλη η εξή προσέγγιση. Πως θέλουμε μια καλή πολιτική συνοχής για τους πολίτες, για τις περιφέρειες, για τους Δήμους και εάν μπορέσουμε να το κλείσουμε και πούμε πως έχουμε μια συμφωνία, τότε νομίζω πως αυτό θα είναι θετικό για όλες τις ε, πλευρές. Βεβαίως ε, δεν μπορώ και να σας ε, διηγηθώ όλα όσα πετύχαμε γιατί υπάρχει το στρες των προηγούμενων εβδομάδων και η κούραση αλλά νομίζω πως το μήνυμα έτσι για το τέλος ε, του έτους είναι θετικό και μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες ε, στις περιφέρειες να γίνει η προετοιμασία για τα επιχειρησιακά προγράμματα, για την εφαρμογή της μελλοντικής πολιτικής συνοχής και βέως με την συμπερίληψη των εταίρων και με τρόπο διάφανο. Και θεωρώ πως ε, αυτούς τους δύσκολους καιρούς το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε και να δείξουμε πως τα έξω είναι αυτό. Και αναγνωρίζεται νομίζω πως ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα θεσμικά όργανα δεν είμαστε μόνο μαζεμένοι γραφειοκράτες αλλά ασχολούμαστε και με τον κόσμο, με τους ανθρώπους και προσπαθούμε να τους ε, στηρίξουμε. Γι' αυτό πρέπει νομίζω να πούμε πως ε, είναι σημαντικό και για τις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις και ελπίζω η Ιρλανδική Προεδρία να το κάνει γιατί το συνέδεσε ούτως ή άλλως η Κυπριακή Προεδρία πως θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να προχωρήσουμε με τρόπο διάφανο και μετά τους τρεις-τέσσερις ε, τριμερείς ε, διαλόγους νομίζω πως είχαμε κάποια δυναμική. Γι' αυτό το οποίο είπε τώρα ο Λάμπερτ για τις μουσιονομικές προοπτικές δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Η όλη αυτή η διαδικασία των δομών στην πολιτική συνοχή βεβαίως έχει μόνο νόημα αν υπάρχει και η αναγκαία χρηματοδότηση και αυτό δεν έχει γίνει και ανησυχώ ιδιαίτερα για το τι θα μπορούσε να προκύψει. κάποια στιγμή θα πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες του το Κοινοβούλιο, αλλά ακόμα ε, ελπίζω πως πρώτον δεν θα καταστραφεί ο κόσμος 21 Δεκεμβρίου και δεύτερον θα υπάρξει συμφωνία για το δημοσιονομικό πλαίσιο με τα κράτη-μέλη και νομίζω πως έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε τη μετάβαση από τη μία προεδρία στην άλλη. Και ελπίζω η συνεργασία να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν ήμουν εγώ παρόν στον ε, τριμέρι διάλογο όπως η Κωστός και ο Λάμπερτ. Γι' αυτό σας αφήσω να απαντήσετε στις παρατηρήσεις που έκανε εκείνη. Απλώς θα ήθελα να πω ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή να αρχίζει να τίθεται σε διαδικασία μια νέα διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή λοιπόν την νεοτεριστική, αν θέλετε, την καινοτόμο κατάσταση, την άρχισε η Κυπριακή Προεδρία. Επιτέλεσε πολύ σημαντική δουλειά. Θα ήθελα να τονίσω το εξή. Παρά το γεγονό ότι υπήρχε τρομερό φόρτο εργασία και πάρα πολλέ ήταν οι ευθύνε τη Κυπριακή Προεδρία, κατορθώσατε το Συμβούλιο να λάβει υπόψη αυτή την μακροπεριφερειακή ε, στρατηγική, αρχίζοντας από την Μεσόγειο. Θα ήθελα λοιπόν αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική πρόοδος να το επισημάνω και να πω ότι ήταν κάτι το πολύ... Δεν ξέρω κύριε Υπουργέ αν θέλετε να απαντήσετε τώρα ή αν θέλετε. Απαντάτε και μετά ακούω στους άλλους συναδέλφους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη ευχαρίστηση σας ευχαριστώ πολύ για τις πάρα πολύ επικοδομητικές παρατηρήσεις και σχόλια που κάνατε. Όπως είπατε, από την αρχή της εφαρμογής της συνθήκης Λισαβόνας οδηγούμεθα σε νέο δρόμο. Τον διανύουμε τώρα. Πρόκειται για μια νέα διαδικασία. Όντω δεν υπήρχε πρώτερη εμπειρία. Είναι πρώτη φορά που τα κράτη-μέλη και οι αρχές γνωρίζουν πλέον την συνήθεια αυτή η νομοθετική διαδικασία, την συναπόφαση, όλοι μαθαίνουμε, ακόμη και οι εθνικές και περιφερειακές αρχές. Όλοι, όλοι μέσα αυτή τη διαδικασία μαθαίνουμε. Βεβαίως, όταν πήραμε την Προεδρία, πρέπει να πω ότι ανακαλύψαμε ότι υπήρχαν πάρα πολλές εντάσεις, πολύ στρες. Ο καθένας προσπαθούσε να ορίσει και να οριοθετήσει το δικό του πεδίο. Από ηθική πλευρά, λοιπόν, θα πρέπει οποιαδήποτε αντιπαράθεση να αποφευχθεί Και αυτή εξ αρχή συνειδητοποίησαμε ότι ο μόνο τρόπο που είχαμε για να προοδεύσουν ήταν να συνεργαστούμε σύμφωνα με τις συνθήκες, σεβόμενες ο καθένας τα προνόμια και τις εξουσίες του καθενός. με πλήρη διαφάνεια, με πλήρη σεβασμό προς τα άτομα και τις αρχές τους, τις αρχές του καθενός. Το είπα πολλές φορές ότι αυτό το οποίο θέλαμε εμείς είναι να μπορέσουν άτομα και οι θεσμοί καλή την πίστη να γνωριστούν και να επικοινωνούν μαζί του. Αν λοιπόν ήταν έστω και μικρή η συνεισφορά μας προς αυτή την κατεύθυνση, Χαίρομαι ιδιαίτερο και χαίρομαι διότι φαίνεται ότι όλοι εκτιμάτε τις προσπάθειες που καταβάλαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Βαρνίστερ Λόι, σωστά. Μιλήσατε για το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει και πάλι πρόκειται για θεσμικό πρόβλημα. Δηλαδή, στοιχεία τα οποία εισήχθησαν στο πολιετές και τα οποία δεν συζητήθηκαν τη διάρκεια των τομεακών διαπραγματεύσεων. Ο νόμος τρόπος που βρήκαμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό είναι να πούμε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο προδικάζει τις αποφάσεις που ληφθούν στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης και παρά το γεγονό ότι αντιστρέψαν κάποιοι, κάποια πράγματα, το ότι μπορέσαμε τελικά να καταλήξουμε στα πλαίσια του πολιετούς σε κάποια συμφωνία είναι κάτι θετικό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το είδαμε και στι δικέ και είναι ένα τρόπο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα από τη δική σα πλευρά. Διότι το Συμβούλιο μα λέει, τα συμπεριλάβαμε αυτά τα στοιχεία, δεν πήραμε τίποτε, δεν το αφαιρέσαμε από τη φωνία, διότι είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την σφαιρική συμφωνία που θα κάνουμε. Αν θέλετε λοιπόν, αυτό ήταν ο καλύτερο τρόπο που βρήκαμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Τώρα, όσον αφορά τα σχόλια τη κυρία Κέλ. Σα ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την συνεισφορά σα. Όλοι γνωρίζουμε πόσα πολλά κάνατε. Και επίσης γνωρίζουμε ότι κατά κάποιο τρόπο είστε η νονά των ε, θεμάτων αυτών για τις επενδύσεις και τα δραστηριότητα και τα διαθετικά ταμεία. Ελπίζουμε ότι τελικά αυτή η νέα δυναμική που δημιουργήθηκε θα μας βοηθήσει να έχουμε μια πραγματικά αποδοτική πολιτική συνοχή. Και αυτά που είπατε και εσείς και ο κύριος Βαρνίστερ όντως πρέπει να πω ότι υπάρχει στο πολιοτές ε, μείωση, περικοπές, δεν μπορέσαμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε την πολιτική συνοχής και να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις των περικοπών στο πλαίσιο του ε, δυνατού. Χωρίς να θέλω να είμαι περισσιόδοξος, κατά την άποψή μου, νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία, αλλά η συμφωνία αυτή θα απαιτήσει αύξηση των κονδυλίων που πηγαίνουν στην συνοχή. Αυτά βλέπω, αυτά ελπίζω ότι θα συμβούν. Θα δούμε στην πραγματικότητα τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Δεν είμαι όμως απεσιόδοξο. δεν είμαι πολύ απεσιόδοξος. Τώρα, σε σχέση με την ερωτήσει του κυρίου Αλφονσί, σωστά, επισήμανε ότι όπως είπαμε, πρόκειται για μια νέα διαδικασία, τη δοκιμάζουμε σιγά σιγά, Όντως είναι νέα διαδικασία, διαδικασία την οποία τη γνωρίζουμε εδώ και ε, τρία χρόνια στα πλαίσια της Συνήξης Λισαβόνας. Πρώτη φορά την εφαρμόζουμε και όπως σας είπα, σιγά σιγά ελπίζω ότι θα, κάνουμε, θα την ε, προχωρήσουμε σωστά. Και σας λέω επίσης ότι στα πλαίσια αυτών που είπατε, στα πλαίσια της μακροστρατηγικής, ε, μακροπεριφερικής στρατηγικής για τη Μεσόγειο θα έχουμε καλές, ε, καλά αποτελέσματα. Βλάσακ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την ε, συνεργασία που είχαμε. Βεβαίως, ε, στην αρχή ξεκινήσαμε λίγο αργά, αλλά χάρη στους πιο έμπειρους ε, συναδέλφους μας προχωρήσαμε στο προπαρασκευαστικό μας ε, έργο. Προχωρήσαμε γρήγορα πριν ε, τις καλοκαιρινές διακοπές. Διαλέξαμε τους πιο έμπειρους ε, συναδέλφους στην διαπραγματευτική ομάδα. Εγώ δεν ήμουν στην πρώτη γραμμή, αλλά συμμετείχα και στους πέντε τριμερείς διαλόγους και μετά από κάποιο διστακτικό ξεκίνημα νομίζω πως είχαμε επιτύχει μεγάλη πρόοδο. Αλλά έχω ένα αίτημα προς εσάς κύριε Υπουργέ, γιατί νομίζω πως ε, η περίοδος αυτή του δισταγμού κράτησε πολύ όταν προσπαθούσαμε δηλαδή να δούμε τι σκόπευε να κάνει ο καθένας ε, από εμάς. Δεν θέλω να επαναληφθούν αυτά όταν θα έχουμε την Ιρλανδική Προεδρία. Ε, δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο και πρέπει να εγκρίνουμε τους κανονισμούς αυτούς το συντομότερο δυνατόν. αλλιώ. θα έχουμε προβλήματα για να αντληθούν οι πόροι. Σας παρακαλώ λοιπόν να διαβάσετε αυτή την εμπειρία στην Ιρλανδική Προεδρία για να συνεχιστεί ε, πρόσκοπτα η συνεργασία. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους γιατί ξέρω πως ήταν ε, επίπονες ε, και απαιτητικέ οι διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Σε μαρζή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα για τις πολιετές. Αφενός και για τον γενικό ρεσμό. Εξ ονόματος ομάδας μου πρώτα απ' όλα της Αττικής Αριστεράς θα ήθελα να χαιρετήσω την εργασία που επιτέλεσε η Κυπριακή Προεδρία στα πλαίσια της Προεδρίας σας πρέπει να πω ότι διαδραματίσατε σημαντικό ρόλο μεταξύ των φίλων της συνοχής και πιστεύω ότι η εργασία σας επέτρεψε να βελτιωθεί η τελευταία πρόταση που υπέβαλε ο πρόεδρος Βον Ρομπάι. Ξέρουμε ότι χωρίς την συνδρομή των φίλων της συνοχής και χωρίς το ρόλο που διαδραμάτισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα είμαστε, όπως είπατε και εσείς εξάλλου, τόσο αισιόδοξοι όσο μπορούμε να είμαστε σήμερα, παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι προσανατολιζόμαστε προς μία γενικότερη μείωση των πιστώσεων που δίδονται στην πολιτική συνοχή. Αυτό είναι ένα προηγούμενο στην ε, ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι για πρώτη φορά η πολιτική συνοχής θα καταγράψει μείωση των κονδυλίων. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι αναλάβατε σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυτή την Προεδρία. Εξαιτίας πρώτα απ' όλα της κρίσης που βαρύνει τους πάντες και τα πάντα και κυρίως εξαιτία της θέσης κάποιων κρατών μελών, των πιο πλουσίων, αυτών που θέλουν ε, να ξοδεύουν τα περισσότερα ή καλύτερα να ξοδεύουμε, που έφτασαν στο Συμβούλιο προτάσσοντας εθνικά συμφέροντα αντί να μιλούν για το γενικότερο ευρωπαϊκό συμφέρον. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπάθησε ιδιαίτερα να τονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άρα το έργο, το δικό σας ως Προεδρία δεν ήταν εύκολο και ειλικρινά και πάλι θα ήθελα να υπογραμμίσω την ποιότητα της εργασίας την οποία επιτελέσατε, ελπίζοντας ότι και η επόμενη Προεδρία, η Ιρλανδική, θα συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση. Ούτως ή άλλως γνωρίζω ότι η δική σας η Προεδρία στο Συμβούλιο θα είναι πάντα μια προσφυλής προεδρία για τους φίλους της συνοχής, διότι θέλουμε να προστατεύονται όλες οι ενδέστερες ε, περιοχές της Ευρώπης από τις περικοπές και τα προβλήματα. Εγώ ήμουν μέλος της ομάδας διαπραγμάτευσης και πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή είμαι σε μια κάπως ιδιότυπη κατάσταση διότι χρειάστηκε να αρχίσουμε την διαπραγμάτευση ενώ δεν ξέραμε ακόμη ποιο είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό όμως δεν μας εμπόδισε να καταλήξουμε σε αποφάσεις για ένα μπλοκ και πρέπει να πω ότι έτσι υλοποίησαμε τους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει. Εξ αρχής να ολοκληρώσουμε δηλαδή τις διαπραγματεύσεις μας πριν από το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω εξ ονόματο τη πολιτικής μου ομάδα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ, Ιωάχιμ Μτσέλλερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ. Εγώ βλέπω κάπως πιο ε, κριτικά τα γεγονότα. Λέτε πως ε, είναι νέα η συνθήκη της Λισαβόνας ε, μα ισχύει ήδη εδώ και τρία χρόνια και πριν ισχύσει είχαμε πολλά χρόνια προετοιμασίας. Οπότε το περιεχόμενο της συνθήκης δεν θα έπρεπε να είναι άγνωστο. Και το ότι το Κοινοβούλιο είναι πλέον στην πλήρη συναπόφαση και για τους ε, τομείς αυτούς ε, ίσχυε και για το ε, και για την περίοδο 2006-2013. Οπότε και αυτό δεν θα έπρεπε να είναι άγνωστο. Και βλέπω εδώ πέρα πως οι προσπάθειες που κατεβαλε ειδικά η Κυπριακή Προεδρία για να προχωρήσει η διαπραγμάτευση είχαν ε, ήταν βεβαίως πάρα πολύ μεγάλες, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι πολύ εντυπωσιακά. βεβαίω δεν, ε, δεν φταίτε εσείς γι' αυτό, έχετε άλλε 26 χώρε με τις οποίες πρέπει να διαπραγματευτείτε. Ε, η Επιτροπή μας τώρα όσον αφορά τον ε, κανονισμό των διαρθρωτικών ταμείων κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη τον Ιούλιο είχαμε εμείς ε, μια βάση για να διαπραγματευτούμε ως ε, κοινοβούλιο και αναφέρθηκε αυτό πως ε, θέλαμε ε, να έχουμε και εμείς μια ίση φωνή. Αλλά... Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συζήτηση των προσχεδίων των κανονισμών πριν οδηγηθούμε σε αποφάσεις. Και υπάρχουν κάποιοι ε, τομείς οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν ε, ιερές ε, αγελάδες και αν δούμε το τι γίνεται και στον προπολογισμό του 2013 και στις διάφορες προτάσεις του Συμβουλίου φαίνεται πως παραμένουν ιερές αγελάδες όπως η Γεωργία ή η Αλληλεία και όταν φτάνουν στην πολιτική την περιφερειακή μιλάνε για αναλογίες και τα λοιπά, παρά το ότι πολλά μέλη του Συμβουλίου πριν από λίγους μήνες όταν τα ρωτούσαν ποιοι είναι οι ευρωπαϊκοί προπολογισμοί με τους οποίους θα επιτύχουμε ανάπτυξη, καινοτομία, επενδύσεις, αμέσως ε, παρέπεμπαν στα διαρθρωτικά ταμεία. Και όταν, λέτε πως, ε, όταν λέγεται πως δεν είναι πολύ αργά να καταλήξουμε συμβασμούς, ναι εντάξει καλώς, αλλά σε λίγες μέρες θα έχουμε 2013 και τελειώνει άρα η τρέχουσα προγραμματική περίοδος και οι περιφέρειες ε, είναι απελπισμένες. Θέλουν να ξεκινήσουν με τα έργα των ε, επιχειρησιακών ε, προγραμμάτων και οι εργασίες δεν μπορούν να ξεκινήσουν γιατί εμείς ασχολούμαστε με τεχνικές ε, λεπτομέρειες ενώ είναι, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα το γενικότερο πλαίσιο και εξαρτάται από το τι χρήματα θα έχουμε τελικά στην ε, διάθεσή μας. Εάν έχουμε δηλαδή ε, μεγάλες περικοπές θα πρέπει να τα ξαναξεκινήσουν όλα από την αρχή αντί να μιλάμε για, για λεπτομέρειες. Κοιτάξτε τώρα... Εγώ είμαι βεβαίως ε, υπεύθυνο ε, για την ε, περιφερειακή συνοχή και θα έπρεπε εκεί πέρα να έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα γρηγορότερα σε σχέση με άλλους κανονισμούς οι οποίοι εξαρτώνται από το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Βέβαια, ε, ήταν θετικές οι επαφές με την Προεδρία του Συμβουλίου και ελπίζω στο επόμενο εξάμεινο να μπορέσουμε να καταλήξουμε όσον αφορά την εδαφική συνοχή. Τώρα, ε, ελπίζω πως θα συνεχίσετε να είστε στο πλευρό μας εντός του Συμβουλίου για τη σημασία της περιφερειακής πολιτικής για να μην χαθεί το θέμα αυτό και υποθέτω πως αν ε, ε, φύγουν 70 ε, δισεκατομμύρια από τον τομέα αυτόν όπως ζητάει Κομισιόν και Κοινοβούλιο μιλάμε για ένα Μιλάμε για άλλους προϋπολογισμούς ε, που έχουν ένα σύμπλην 5 δισεκατομμυρίων από το ένα έτος ε, στο, άλλο. Και ειδικά σκεφτούμε το τι γίνεται στα κράτη-μέλη, δεν αντιλαμβάνομαι πλέον πλήρως την ε, κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσει ένα αποφασιστικό βήμα το Συμβούλιο και να μπορέσει έτσι να χρηματοδοτήσει την ε, πολιτική ε, συνοχής καθώς είναι από τα κύρια αναπτυξιακά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννη Ολμπριχτ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ε, είχα θετικές εμπειρίες από τον τριμερή διάλογο. και ούτως ή άλλως τα πράγματα συνεχίζονται. Έχω δύο ερωτήσεις, οι οποίες δεν είναι πολύ διπλωματικές, αλλά πώς βλέπετε εσείς ε, ως ε, μέλος ε, του Συμβουλίου την θέση των κρατών μελών σήμερα, στο τέλος του 2012, απέναντι στην πολιτική συνοχής καθώς στην προετοιμασία του διαλόγου βεβαίως είχατε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε με τα κράτη-μέλη και πολύ ορθά ε, δεν ε, εκφράσατε τη θέση της, ε, της Κύπρου. Οπότε όταν θα επανέλθετε ως ένα απλό μέλος του Συμβουλίου, ποια θα είναι η θέση της Κύπρου, θα είστε φίλος συνοχής ή φίλος των καλύτερων δαπανών. Ελίζα Μπερσέτλε. Ναι, μα αυτό ακριβώς είναι το θέμα, Γιάν. Πρέπει να πω πως ναι, πράγματι η Κυπριακή Προεδρία πιθανώς έζησε ως πρώτη Προεδρία το τι σημαίνει συναπόφαση στον τομέα αυτών, δηλαδή Μέχρι τώρα είχαμε τη λεγόμενη μέθοδο του Βερολίνου, έστελναν επιστολές και έκαναν ό,τι θέλανε. Αυτές οι εποχές τελείωσαν. Και χρειάστηκε χρόνος για να το αντιληφθεί αυτό το Συμβούλιο. Αλλά νομίζω πως ο τελευταίος μήνας ήταν επιτυχής ε, σε πολλούς τομείς. Ε, τουλάχιστον η διαπραγματευτική βάση ήταν καλύτερη από ό,τι πιο πριν και αυτό νομίζω ήταν σημαντικό το ότι αναγνωριστήκαμε δηλαδή ως ισότιμη εταίροι. Βεβαίως είναι σαφές πως θέλουμε μια διάφανη και αποτελεσματική διαρθρωτική πολιτική. Τονίζω το διάφανη. Αν έχετε τη δυνατότητα να το πείτε κάτι μέλη θα ήταν θετικό και Θα επιμείνουμε σε αυτό και βέβαια είναι δύσκολο να θεωρούμε πως μπορούμε να συνεχίσουμε όπως τώρα. Και αυτό νομίζω είναι η μεγάλη δυσκολία. Η Προεδρία του Συμβουλίου είχε ακριβώς πάντα το πρόβλημα α, της ε, διαμεσολάβησης μεταξύ των κρατών μελών που θεωρούσαν πως τα πράγματα μπορούν να συνεχίσουν όπως είχαν και του Κοινοβουλίου που είχε την αντίθετη άποψη. Και εκεί πέρα Νομίζω θα πρέπει αυτό να συνεχίσετε να το κάνετε και τις επόμενες μέρες, το μεσολαβητικό αυτό ρόλο δηλαδή, και νομίζω πως ε, δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι στο Συμβούλιο και αυτό δεν είναι κριτική σε εσά, αλλά στο Συμβούλιο, πως χρειάζεται και ε, να αποκτήσει αυτές τις διοικητικές ικανότητες ε, το Συμβούλιο, κάτι το οποίο συχνά συζητάμε. Και αυτό πρέπει να το δώσετε ως μήνυμα και στην Ιρλανδέζικη Προεδρία. Δηλαδή, οι διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν μόνο αν γίνονται ε, παράλληλα και όχι άμα κάθεται ε, χωρίς, ε, άμα είναι τελείως αμετακίνητο το Συμβούλιο. Αυτή την εμπειρία πρέπει να μεταδώσετε στο Συμβούλιο. Κάτι τελευταίο. Το ζήτημα του και το τι είναι εκεί πέρα το αντικείμενο διαπραγμάτευση. Έχω το πρόβλημα πως πάλι ακολουθείται η μέθοδος Βερολίνου. Και δεν αντιλαμβάνομαι πως θα έχουμε ένα αποτέλεσμα του πολιτικού δημοσιονομικού πλησίου γιατί ήμουν παρούσα και το θυμάμαι. Δηλαδή, ήταν μια τεράστια λίστα αυτή η οποία είχε έρθει. Μα δεν θα είχαμε τελειώσει με τις ε, διαπραγματεύσεις ε, με τους ε, μεγάλους κανονισμούς. Και μόλις έφυγε από τον κανονικό, από τον κανονισμό πλαίσιο και πήγε στο Πουδουπού, είδαμε πως δεν ήταν οι αποφασιστικές ε, παράγραφοι έτοιμες γιατί πλέον δεν τέριαζαν σε ένα προετοιμασμένο συνεκτικό έγγραφο. Και ε, ξού και οι εκκλήσεις ε, στις τελευταίες διαπραγματεύσεις πως πράγματα τα οποία είναι στον κανονισμό πλαίσιο δεν μπορούν να πάνε στο Πουδουπού. Υπάρχουν ε, εντάξει, πράγματα που συζητιούνται, αλλά όχι. Δεν μιλούσαν για κανόνα κανόνα, αναβολές, ε, για τα ποσοστά της 100. Κάποιοι ήθελαν να διατηρήσουν, όπως είπα, τη μέθοδο του Βερολίνου, η οποία, όπως σας είπα, δεν, δεν υπάρχει πια. Δεν είναι αυτή η διαπραγμάτευση. Το Κοινοβούλιο θέλει μια συνεκτική πολιτική. Γιατί αυτό ακριβώς είναι η πρόοδος. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, χωρίς να κάνω περαιτέρω παρατηρήσεις και να πω ευγενικά πράγματα. Θα σας ευχαριστήσω για τον τριμερή διάλογο, διότι μπορέσετε με την ομάδα σας να κάνετε πολύ καλή διαπραγμάτευση. Δεύτερον, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον πολύ σωστό και θετικό τρόπο που ε, αντιμετωπίσατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνυπεύθυνο για θέματα της δικής θερμοκρατίας. Οι άλλοι θα ακολουθήσουν το δικό σας παράδειγμα. Θα ήθελα να πω ότι αφήνετε ένα μεγάλο και σημαντικό κληροδότημα το οποίο θα πρέπει να περάσει στην επόμενη Προεδρία, διότι για μας, για την Επιτροπή μας, αυτή είναι η προτεραιότητα των προτεραιοτήτων. Να περάσει το μήνυμα και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας περαιτέρω για να καταλήξουμε σε συμβαστική ε, λύση. Derek Vaughan, επόμενος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στον Υπουργό ότι χαιρόμαστε που τον βλέπουμε σε μια συνεδρίαση στην οποία δεν έχει να κάνει με χρήμα και με διαπραγματεύσει του προπολογισμού. Πολλές φορές συναντηθήκαμε τους τελευταίους μήνες και εβδομάδες. Σήμερα εστιαζόμαστε στο επόμενο MFF, στο επόμενο Αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό το 6-12 και τον 13, ε, διότι του χρόνου θα είναι το τελευταίο έτος του παρόντος πολιετούς ε, πλαισίου δημοσιονομικών προπτικών. Και ξέρω ότι δεν ήταν εύκολα ε, ό,τι έγινε για να καταλήξουμε και για τον διορθωτικό, τον φετινό προϋπολογισμό και του χρόνου ε, τα πράγματα. Πολύ σωστά το χειριστήκατε. Σύμφωνα με την Επιτροπή θα μας λείπουν 9 ε, δις για του χρόνου. Τρία εφέτος και έξι του χρόνου ίσως. Τα πρώτα τρία δις φαίνεται ότι ε, πέφτουν ε, στον κλήρο της ε, πολιτικής συνοχής. Πράγμα το οποίο επίσης θα επηρεάσει την κατάσταση του χρόνου. Τελειώνοντας σήμερα μπορούσατε να μας πείτε λίγο πιο... Έτσι, με πιο ελαφρύ πράγμα. Πιστεύετε ότι το Συμβούλιο θα δεχθεί να υπάρχει για φέτος αυτό το πρόβλημα των τριών δίσκων με τον προπολογισμό και του χρόνου το επίσης. Επίσης, πόσα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα επηρεαστούν του χρόνου στα πλαίσια της πολιτικής ε, συνεχής. Ε, διότι πιστεύουμε ότι αυτό το πρόβλημα εμείς στο Κοινοβούλιο θα δημιουργήσει πρόβλημα, διότι κάποιες ε, ε δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν και από νομική πλευρά επίση έχουμε πρόβλημα. Και τελειώνουμε με ελληνικά, με τον κύριο Αγκουράκη και μετά με τον κύριο Σταυρακάκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν θέλετε μπορώ και σε γερμανικά, αλλά προτιμώ τα ελληνικά, έχετε δίκιο. Καταρχήν ε, να σας ευχηθώ ότι καλύτερο κύριε Υπουργέ και καλές γιορτές. Ε, Δύο-τρεις παρατηρήσεις στα όσα είπατε. Ε, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ε, θέλω να μεταφέρω σε αυτή την αίθουσα την αγωνία χιλιάδων εργαζομένων στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση οι οποίοι εδώ και εβδομάδες είναι σε μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις διότι απειλείται η ύπαρξή τους, στην ουσία βρίσκονται στο δρόμο απολυμμένοι, εντελώς άδικα και αυτό καταλαβαίνετε δημιουργεί τεράστια προβλήματα και δείχνει ε, πού βρισκόμαστε σήμερα. Δεν είναι τυχαία που επέλεξα αυτό το στοιχείο για, να, για την τοποθέτησή μου. Γιατί αντίθετα με άλλους ε, αξιότιμους ε, βουλευτές που πήραν το λόγο, προσωπικά πιστεύω ότι τα προβλήματα που είχατε στο Συμβούλιο δεν ήταν τόσο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου, αλλά το πρόβλημα το μεγάλο ήταν ότι υπάρχουν μεγάλοι ανταγωνισμοί, μεγάλες διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό φυσικά είναι αποτέλεσμα της κρίσης. Η κρίση δυστυχώς θα ενταθεί το επόμενο χρόνο και μετά και άρα αυτές οι αντιπαραθέσεις θα οξύνονται και θα αντιπαρατίθενται ακόμα πιο πολύ. Δεν πιστεύω ότι δηλαδή το θέμα είναι better spending. Το πρόβλημα είναι less spending, να το πω έτσι ξεκάθαρα, διότι είναι η κρίση. Σε σχέση με αυτό κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι θεωρώ, χωρίς να σημαίνει ότι εγκαλώ εσάς ή την ε, ε, Κυπριακή Προεδρία, πάντως, αν κατάλαβα καλά, ε, είπατε ότι ε, από εδώ και στο εξή, στα πλαίσια του εξαμήνου και στα πλαίσια της ενισχυμένης διακυβέρνησης, θα γίνεται μια συλλογική ανασκόπηση, θεώρηση, δεν, δεν κατάλαβα ακριβώς, της πολιτικής συνοχής. Εάν αυτό τώρα το κατάλαβα σωστά και με τα δεδομένα που ξέρω μέχρι τώρα, αυτό σημαίνει εξάμεινο και ενισχυμένη διακυβέρνηση περικοπές. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν. Είναι οι γνωστές conditionalities. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω γύρω από το ζήτημα αυτό. Και τέλος, δυστυχώς και σήμερα βέβαια η συζήτηση ε, περιστράφηκε στα, στο ύψος των ποσών, η οποία έχει τη σημασία της, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Εν ε, νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι τα ποσά αυτά ε, δεν έχουν σχέση με πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, που η κρίση οξύνει ακόμα περισσότερο αυτές τις ανάγκες και εννοώ απασχόληση, ενώ εκπαίδευση ποιότητας, ενώ ανθρώπινες συνθήκες ζωής στις πόλεις έστω και αυτά τα ποσά κατευθύνονται στο μεγάλο μονοπωλιακό κεφάλαιο το οποίο αναζητά τρόπους φθηνού χρήματο μπροστά σε συνθήκε τη κρίση. Και από αυτή την άποψη, επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι σχεδόν βέβαιο ότι και τα ποσά αυτά όχι απλώ δεν θα συμβάλλουν στη συνοχή, αλλά αντίθετα θα συμβάλλουν σε ακόμα μεγαλύτερη απόκληση και σε ακόμα περισσότερα κοινωνικά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσά και στον Κυπριακό λαό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Ε, δεν σας κρύβω ένα γεγονό που πραγματικά το ζήσαμε πάρα πολλοί συνάδελφοι. Ε, την ε, Πριν η Κυπριακή Δημοκρατία αναλάβει την Προεδρία, είχαν εκφραστεί κάποιες ανησυχίες πώς είναι δυνατόν μια μικρή χώρα να μπορεί να διαπραγματευτεί τόσο δύσκολα προβλήματα όπως ήταν ο προπολογισμό, το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, κανονισμοί και τόσα άρα δύσκολα προβλήματα μεσούς της οικονομικής κρίσης. Αποδείξατε λοιπόν ότι με τις προσπάθειες και με την ικανότητα που χειριστήκατε και διαπραγματευτήκατε τα θέματα ότι και μια πολύ μικρή χώρα μπορεί να έχει μια πολύ καλή και αποτελεσματική προεδρία. Ε, σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο και για σας και για τον Κυπριακό λαό. Okay, thank you, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για τις ε, πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις με τη σειρά. Ενδεχομένως βέβαια κάποιες απαντήσεις να φέρονται σε περισσότερες από μία ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι χρειάζεται μία συνέχεια και θα πρέπει να καταφέρουμε ομαλά να περάσουμε στην Ιρλανδική Προεδρία όλη αυτή την εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει και θα πρέπει να συνεχίσουμε στο δρόμο αυτό προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό. Επομένως, ε, πραγματικά και εγώ και οι συναδελφοί μου δεσμευόμαστε προκειμένου να συνεργαστούμε αμέσως τις επόμενες μάλιστα ημέρες με την Ιρλανδική Προεδρία. Ξέρετε ότι τις τελευταίες έξι εβδομάδες ήταν και αυτοί παρόντες, συνεργάζονταν μαζί μας προκειμένου να εξασφαλίσουν ακριβώς αυτό, μια ομαλή διαβίβαση στη δική τους ε, Προεδρία. Θέλουμε να πετύχουμε συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι και οι Ιρλανδοί θα συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο με εμά. Όσον αφορά τώρα τις ε, επόμενε ερωτήσεις του κ. Αλφονσί. Νομίζω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταβληθεί μια σημαντική συνεχής προσπάθεια προκειμένου να καταφέρουμε να προστατεύσουμε την πολιτική συνοχής. Όντω, αληθεύει ότι όπω όλε οι υπόλοιπε κοινωνικέ πολιτικέ δέχεται έντονη πίεση αυτή τη στιγμή. Εμείς ε, ως ειλικρινείς διαμεσολαβητές έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση και τη δημοσιονομική των κρατών μελών. Δεν ήταν η επιλογή μας αυτή, δεν μας άρεσε κάτι τέτοιο, αλλά ήταν αναπόφευκτο να κάνουμε κάποιες προτάσεις μείωσης, περικοπής, που επηρεάζουν όλα τα τμήματα και τα υποτμήματα της πολιτικής αυτής. Προσπαθήσαμε πάντως στο μέτρο του δυνατού κάθε φορά να διατηρήσουμε την πολιτική συνοχής και να διατηρήσουμε πάλι στο μέτρο του δυνατού την υποστήριξη προς τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Αν υπάρχει μάλιστα ένα σημείο επί του οποίου υπήρχε μια γενικότερη συμφωνία και απαντώ κατά αυτόν τον τρόπο και στην ερώτηση που έθεσε ο κύριος Όλμπριχτ, αν υπάρχει, επαναλαμβάνω, κάποιο σημείο επί του οποίου τα κράτη-μέλη βλέπαν τα πράγματα με έναν τρόπο λίγο πιο συνενετικό, το σημείο αυτό είναι η αναγκαιότητα να επικεντρωθεί η πολιτική συνοχή στις λιγότερο προηγμένες περιφέρειες. Θετικό λοιπόν αυτό. Ξέρουμε όλοι ότι από μόνο του δεν αρκεί, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε όλα τα επιμέρους τμήματα της πολιτικής συνοχής. Η έμφαση όμως που δόθηκε στις λιγότερα αναπτυγμένες περιφέρειες θεωρώταν μια θετική εξέλιξη. Εν συνεχεία, γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει αυτή η αέναη διαπραγμάτευση, αντιπαράθεση ανάμεσα στα όσα γίνονται σε επίπεδο τεχνολογίας, σε ό,τι αφορά δηλαδή την πολιτική του μέλλοντος και σε αυτό το οποίο γίνεται σε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι οι χώρες εκείνες οι οποίες εποφελούνται από τα προγράμματα τεχνολογίας, από την έρευνα, τελικά είναι ελάχιστε. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να εμπλέξουμε όλα τα κράτη-μέλη και να καταφέρουμε να βρούμε τη μέγιστη δυνατή διασύνδεση ανάμεσα στην αριστεία που θα πρέπει βέβαια να χαρακτηρίζει ένα πρόγραμμα έρευνας και από την άλλη ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε κλιμάκωση της αριστείας στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Δεν θα πρέπει χρησιμοποιώντας την επιστημονική αριστεία ως πρόσχημα να αποκλείουμε ολόκληρα κράτη-μέλη από τα ωφέλη της έρευνας και της τεχνολογίας. Προσπαθήσαμε λοιπόν πάλι στο μέτρο του δυνατού να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή διάρθρωση ανάμεσα στις δύο αυτές διαστάσεις. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις ε, του κυρίου Ζέλερ, ξέρετε, έχετε απόλυτο δίκιο στις επικρίσεις τις οποίες εκφράσατε. Συμφωνώ ότι ήταν αναπόφευκτες οι περικοπές, οι μειώσεις ε, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεδομένων βέβαια και των θέσεων των βασικών κρατών μελών που συμβάλλουν στον κοινοτικό προπολογισμό. Αν έχετε κάποια κράτη-μέλη τα οποία συμβάλλουν στον προπολογισμό πάνω από τα δύο τρίτα και που τελικά εκπροσωπούν περισσότερο από το ίμιση του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία ζητάνε συνεχώς μειώσεις, ε, δεν μπορείτε να τα γνωρίσετε αυτά τα κράτη-μέλη. Πρέπει κατά κάποιο τρόπο να τα εμπλέξετε στην όλη διαδικασία και να καταφέρετε να τα πείσετε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και βεβαίως ε, δεν συμφωνώ με την ιδέα αυτή την οποία την έφερε και ο κύριος Όλμπρικτ, ότι η καλύτερη χρησιμοποίηση των πόρων σημαίνει ουσιαστικά λιγότερη πόρη. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι αντί να μιλάμε με δεδομένα μικρότερων διαθέσιμων πόρων, να μιλάμε καλύτερα για την ποιότητα της δαπάνησης των πόρων. Και πιστεύω ότι όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον κάνουμε προσπάθειες προκειμένου τα διαθέσιμα κονδύλια να δαπανώνται πιο ποιοτικά. Και πιστεύω ότι εν τέλει θα καταφέρουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου θα έχουμε μια λύση που θα είναι γενικότερα αποδεκτή από τους καθαρούς εισφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από τη νομική της διάρθρωση, έχει τρεις παράλληλους πυλώνες. Σαφώς έχουμε τα ζητήματα της κοινή αγοράς, αλλά έχουμε επίσης και την συνοχή και την κοινή γεωργική πολιτική. Και ανάμεσα στους τρεις αυτούς πυλώνες υπάρχει μια έντονη διασύνδεση. Και σε οτιδήποτε τελικά κάνουμε, οποιαδήποτε συμφωνία και προσπαθούμε να πετύχουμε, θα πρέπει να μην στρεβλώνουμε την ισορροπία αυτή, προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα αποτελεί πρόοδο όσον αφορά την βελτίωση των επενδύσεων που κάνουμε για το μέλλον και έχοντας κατά νου πάντα βέβαια και την κοινωνική διάσταση, η οποία είναι αναγκαία. Δεν ξεχνάμε ότι ήδη τη δεκαετία του 50, όταν δημιουργήθηκε η κοινή αγορά, η κοινή γεωργική πολιτική τότε, αποτελούσε ήδη τότε την άλλη διάσταση, η οποία τελικά θα αντιστάθμιζε την κοινή αγορά, μέσω μιας πολιτικής που είχε μια καθαρά κοινωνική πτυχή. Τη δεκαετία του 80 δημιουργήσαμε μια γνήσια κοινωνική πολιτική, προκειμένου να αντισταθμίσουμε την έλλειψη συνοχής ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να καταλήξουμε κάποια στιγμή στο σωστό μείγμα πολιτικών. Όσον αφορά τώρα την παρέμβαση του κυρίου Όλμπριχτ. Ξέρετε ότι πολλές φορές οι θέσεις των κρατών μελών, η άποψή τους για την συνοχή, δίσταται πολλές φορές. Από τη μια έχουμε αυτούς που θέλουν ε, καλύτερη χρησιμοποίηση των πόρων που ουσιαστικά θέλουν μείωση του προπολογισμού και πολλά κράτη-μέλη έχουν και διαφορετικές απόψεις. Υπάρχουν ορισμένες χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία ή η Φιλανδία που είναι μέλη αν θέλετε της ομάδας αυτής αλλά παράλληλα θέλουν και μια ισχυρή πολιτική συνοχής και έπειτα στην ομάδα αυτή των κρατών μελών έχουμε ορισμένε που δεν θέλουν μια ισχυρή πολιτική συνοχή, όπω για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιθυμεί μια ισχυρή πολιτική συνοχή. Γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο μα λένε είναι ότι λαμβάνουμε χρήματα στα πλαίσια τη πολιτική συνοχή, τα οποία εμεί δεν θέλουμε. Δεν ακολουθούμε εμεί αυτή την προσέγγιση όσον αφορά τη σχέση μα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμφωνούμε ουσιαστικά με τη στάση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν έχει η κατάσταση, αλλά εν γέννη αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι ε, η πολιτική συνοχής γίνεται ευρύτερα αποδεκτή ακόμη και από τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία δεν συμφωνούν με την πολιτική αυτή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι Δανείοι, ακόμα και πριν να λάβουν την Προεδρία, μας λέγανε δεν μας αρέσει η πολιτική αυτή, αλλά ξέρουμε ότι θα υπάρξει στο μέλλον πολιτική συνοχής, άρα το αποδεχόμαστε ως δεδομένο. Από την άλλη έχουμε και όλα τα κράτη-μέλη που ανήκουν στην ομάδα των φίλων της συνοχής. Είναι 15, με την Κροατία θα γίνουν 16 αυτά τα κράτη-μέλη. Και ξέρετε ότι τα κράτη αυτά επιμένουν πάρα πολύ στο ζήτημα της πολιτικής συνοχής. Παράλληλα, αυτά τα κράτη-μέλη είναι τα πιο αδύναμα από οικονομική πλευρά, όσον αφορά σωστικά την εισφορά του στο κοινοτικό προπολογισμό. Επομένω, δεν μπορούν πραγματικά να πιέσουν για μια ισχυρή πολιτική συνοχή. Σα λέω λοιπόν πάλι ότι θα πρέπει να βρούμε την το κατάλληλο μείγμα πολιτικών. Όσον αφορά τώρα την Κύπρο, η κατάσταση ήταν ιδιάζουσα, γιατί ουσιαστικά οριακά ήμασταν καθαροί φορεί στην αρχή αλλά όλο και περισσότερο πλησιάζαμε το επίπεδο των χωρών συνοχής. Και ως Προεδρία προφανώς δεν μπορούσαμε εμείς να τοποθετηθούμε εθνικά. Συμμετείχαμε σε όλες τις συνεδριάσεις των φίλων της συνοχής, πριν από την Προεδρία μας ως παρατηρητές και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας ως Προεδρεύοντες. Νομίζω πάντως ότι όλοι γνωρίζουν ποια είναι η θέση μας όσον αφορά την πολιτική συνοχής. Προφανώς η Κύπρος θα ταχθεί με τα κράτη-μέλη που ανήκουν στην ομάδα των φίλων της συνοχής. Και όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, και εμείς θέλαμε να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια στην πολιτική συνοχή και να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητε της χώρας μας. Όσον αφορά τα όσα είπε η κυρία Σρέντερ. Έχετε δίκιο ότι πολλέ φορέ προσπαθούμε να συνεχίσουμε με την εργασία μα όπω το παρελθόν, μόλον ότι τα πάντα έχουν τροποποιηθεί. Πιστεύω ωστόσο ότι σιγά σιγά και εμεί προσαρμοζόμαστε και όλο και περισσότεροι τελικά συνειδητοποιούν ότι τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο στο μέλλον, δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο στο μέλλον. Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία ε, αποκόμιση διδαγμάτων για όλου, για όλα τα κράτη-μέλη και αναφέρομαι αυτή τη στιγμή σε έναν τομέα, στον οποίο η Κυπριακή Προεδρία θεωρώ ότι συνέβαλε, γιατί ουσιαστικά αναλάβαμε για πρώτη φορά την Προεδρία, δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένη τοποθέτηση η οποία να βασίζεται σε πρώτερες εμπειρίες μας και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να καταφέρουμε να πετύχουμε μία κάποια πρόοδο, να καταφέρουμε να συμβάλλουμε κι εμείς με το δικό μας το λιθαράκι, προκειμένου να μάθουν τα κράτη-μέλη να λειτουργούν με έναν διαφορετικό τρόπο και να συνεργάζονται με διαφορετικό τρόπο. Εν γέννη, η εμπειρία μας ήταν θετική. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη όντως μαθαίνουν αυτή τη στιγμή και προσαρμόζονται, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξει τελικά η κοινοτροπία τους και η γενικότερη στάση τους. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα θεσμικής φύσης, γιατί όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ξέρετε ότι όσον αφορά το τμήμα των δαπανών, εκεί λαμβάνεται απόφαση του Συμβουλίου αφού δώσει σύμφωνη γνώμη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα, ορισμένα κράτη-μέλη λένε εντάξει, πρόκειται απλώ για μια τυπικότητα, πράγμα το οποίο δεν ισχύει προφανώ. Καταφέραμε λοιπόν το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα να διευθετήσουμε κατά τέτοιο τρόπο τα πράγματα, ώστε να συνεργαστούμε καλύτερα με την ομάδα διαπραγματεύση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσπαθώντα να εξασφαλίσουμε καταρχά ότι λαμβάνονται υπόψη οι γνωμοδοτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεύτερον, ότι ό,τι αποφασιστεί τελικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα έχει εν τέλει και τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρετε ότι όσον αφορά του ιδίου πόρου και όσον αφορά τα έσοδα, εκεί πέρα απαιτείται απόφαση πάλι του Συμβουλίου αφού όμως προηγηθεί μια διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού υπάρξει και έγκριση από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και έπειτα έχουμε και όλες αυτές τις νομοθετικές προτάσεις που εντάσσονται στη συναπόφαση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να συνδέσουμε όλες αυτές τις παραμέτρους. Και κάτι ακόμα που ε, κάνει τα πράγματα ακόμη πιο πολύπλοκα. Το Συμβούλιο διαπραγματεύεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά η τελική πολιτική απόφαση λαμβάνεται σε άλλο επίπεδο, σε επίπεδο αρχηγών, κρατών και κυβερνήσεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει πάλι η σωστή διασύνδεση ανάμεσα στο επίπεδο αυτό των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, το επίπεδο του Συμβουλίου και τη σχέση που θα πρέπει να υπάρχει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε με την συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν είχαμε πρώτερη εμπειρία. Πρέπει λοιπόν εμείς να καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο και σε αυτό. Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Μποστινάρου, σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας και προφανώς θα κάνουμε κάθε τι το δυνατό, δυστυχώς δεν είναι στην αίθουσα ο κύριος Μποστινάρου, θα κάνουμε πάντως κάθε τι το δυνατό προκειμένου να διαβεβάσουμε όλο αυτό το έργο και το πληροδότημα στην Ιρλανδική Προεδρία και να μην χαθεί όλη αυτή η πολύτιμη εμπειρία. Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Βόγκαν, πιστεύω ότι έχουμε συνεργαστεί πολύ θετικά και επικοδομητικά για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας και έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και ότι υπάρχει ένα χάσμα το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί. Προτού να φερθώ σε περισσότερε λεπτομέρειε, πρέπει να σα πω ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε στο Συμβούλιο και κατά την έγκριση τη κοινή τοποθέτηση του Συμβουλίου για τον προπολογισμό 2013, καταφέραμε να έχουμε ένα τίτλο ο οποίο είχε αύξηση, μια γραμμή του προπολογισμού με πολύ σημαντική αύξηση. 2,79% αύξηση για την πολιτική συνοχής ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε περίπου 6%, εμείς καταφέραμε να εξασφαλίσουμε 8,2% αύξηση όσον αφορά τις υποχρώσεις πληρωμών για την πολιτική συνοχή. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό για μας να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε αυτά τα κονδύλια για την πολιτική συνοχή και να αποπληρώσουμε τελικά τους λογαριασμούς, να ανταποκριθούμε ουσιαστικά στι υποχρεώσει μας για την χρηματοδοτική αυτή περίοδο που ολοκληρώνεται και για τις αρχές τη επόμενη χρηματοδοτικής περίοδου. Όσον αφορά τώρα το Συμβούλιο, προφανώς κάθε, κράτο, κάθε κράτος μέλος έχει τις δικές του νομικέ δεσμεύσεις. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά που αναβάλλεται κάτι, εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα. Επίση, υπάρχουν πολλοί στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω να έχουμε πρόσωπο της Επιτροπής που πέρα σήμερα, ότι υπάρχει πάντα δυνατότητα να δοθούν στο μέλλον κάποια χρήματα. Επομένω, κάθε, φορά κάθε φορά έρχονται και μα λένε για ποιο λόγο δεν δίνετε τα χρήματα αυτά σε μια μετέπειτα περίοδο, πάντα θεωρούν ότι είναι δυνατό να μπορούμε να πληρώνουμε χρησιμοποιώντα αποθεματικά προηγούμενων ετών. Πάντως, στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα, και στις δυσκολίες που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε, είδανε πάρα πολλά κράτη-μέλη ότι πολλές φορές έπρεπε να δεσμεύσουν νέα χρήματα προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαι λοιπόν ιδιαίτερα απεσιόδοξο ω προ αυτό. Αυτό μπορώ να σα πω είναι ότι πολλέ φορέ μαθαίνουμε από τα λάθη μα. Ε, δεν, δεν ξέρω κύριε Αγκουράκη τι να πω. Αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις δυσκολίες και υπάρχει όπως είπατε πολύ σωστά μια άμεση σχέση ανάμεσα στις δυσκολίες αυτές και την επίθεση που δέχεται η πολιτική συνοχή. Αναφίβολα υπάρχει μια σχέση και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να προστατεύσουμε τις ε, πληρωμές και να προστατεύσουμε την πολιτική στο σύνολό τη, προσέχοντας ωστόσο να την επικεντρώσουμε με τον σωστό τρόπο. Ε, όπως είπα και προηγουμένως, ε, για μένα το better spending δεν σημαίνει αναγκαστικά λιγότερο spending. Σημαίνει ότι πρέπει να δούμε κάποιες αδυναμίες που υπήρχαν μέχρι τώρα, να τις διορθώσουμε αλλά πρέπει να έχουμε τις σωστές πολιτικές στην υπηρεσία των ε, ε, περιφερειών μας και στην υπηρεσία των ε, αυτών που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη. Όμως αυτό που είπα προηγουμένως δεν αναφερόταν στο, στο θέμα της κατά εξάμεινο αναθεώρησης αν θέλετε. Αυτό που είπα ήταν απλώς η δική μου αίσθηση για το πού θα βρούμε τη συμφωνία για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ότι τελικά, αν θέλετε, στις προσεχείς εβδομάδες για να υπάρξει συμφωνία θα πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο προς τα πάνω, αυτή είναι η δική μου αντίληψη έτσι, την, την χρηματοδότηση της συνοχής. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε επίσης λίγο προς τα πάνω την κοινή αγροτική πολιτική και ενδεχομένως να πρέπει να κάνουμε κάποιες περαιτέρω περικοπές στην ε, ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη και στα μεγάλα προγράμματα. Εκεί βλέπω, αν θέλετε, να βρίσκουμε την συμφωνία. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη από την ε, μέχρι τώρα εμπειρία μου. Ε, τον κύριο Σταυρακάκη δεν έχω να προσθέσω πολλά, απλώς θα ήθελα να τον ευχαριστήσω θερμά και για το ότι ηγήθηκε της αποστολής στην Κύπρο και για όλα όσα έχει κάνει και για τα καλά του λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά. Ε, Madam President. Ε, Κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να τελειώσω με τον ε, σας ευχαριστήσω για όλα όσα έχετε κάνει. Ήταν ευχαρίστηση η συνεργασία μας. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή συνεργασία με την Ιρλανδική Προεδρία. Είναι ικανοί άνθρωποι. Και νομίζω πως ε, πάρα πολύ γρήγορα θα έχουμε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων σας και θα επιτύχουν αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα. Να σας ευχαριστήσω για το Συμβούλιο του Νοεμβρίου, γιατί έλαβε χώρα δύο εβδομάδες πριν από την σημαντική συνοδοκορφή για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και επιλέξατε κάτι το οποίο μας ε, έδωσε την δυνατότητα να στείλουμε το μήνυμα πως έχουμε μια πολιτική επενδύσεων, μια αναπτυξιακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό νομίζω επηρέασε και τις ε, συζητήσεις ε, στις διαπραγματεύσεις πριν από τις συνεδρίες του Συμβουλίου. Και τέλος, βεβαίω έχει δουλειά πρέπει να γίνει ακόμα αυτή τη βδομάδα με τον Αντώνη. Οπότε ελπίζουμε να έχουμε ευτυχές τέλος και να ξεκουραστούμε και τις διακοπές και θα συνεχίσει η Κύπρος να στηρίζει την πολιτική αυτή. Σας ευχαριστώ. Ναι, δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, βεβαίως θα συνεχίσουμε και αυτή τη βδομάδα μέχρι την τελευταία στιγμή και ελπίζω να προχωρήσουμε και θα ήθελα να πω πως εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειες όλων των κρατών μελών για μια επικοδομητική προσέγγιση και νομίζω πως όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε και αυτό το οποίο έχουμε βεβαίω είναι η ναυαρχίδα της επικοδομητικής μας συνεργασίας και εύχομαι σε όλους ε, καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά και καλή συνέχεια στην πολιτική σας. Τώρα να σας ενημερώσω ότι έχουμε την πρώτη μας συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, τον κύριο Βαλτέρ Ντεφά. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Γενικό Διευθυντή και μετά θα έχουμε και χρόνο για ερωτήσεις και σχόλια. Καλώς ήρθατε. Έχετε αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε και χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να εμφανιστώ στην Επιτροπή σας. Όταν ε, διορίστηκα Γενικός ε, Διευθυντής, αμέσως ε, συναντήθηκα με την Πρόεδρο της Επιτροπής σας και τη Γραμματεία έτσι ώστε η γενική μας διεύθυνση να συνεχίζει να σας ε, στηρίζει στο έργο σας. Εγώ τον ξεκίνησα, ο Επίτροπος Χάν ε, μου έδωσε μια ξεκάθαρη αποστολή για το πρώτο έτος. Η αποστολή ήταν η Γενική Διεύθυνση να αρχίσει να λειτουργεί για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ε, προκλήσεις ε, του μέλλοντος. Και οι προκλήσεις είναι πολύ υψηλές. Θα αναφέρω πέντε από αυτές. Η πρώτη είναι να τοποθετηθεί η πολιτική, να καθοριστεί η πολιτική ως μια αναπτυξιακή πολιτική για επενδύσεις και δουλειές με ένα νέο μείγμα οικονομικής πολιτικής που έχει τρία στρώματα. Τρεις, τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι βεβαίως η ε, οικονομική εξυγίανση. Το, δεύτερο διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και το τρίτο σκέλος είναι η ε, στοχευμένες ε, επενδύσεις για την ανάπτυξη και τις δουλειές. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει να τοποθετηθεί η πολιτική. Δεύτερη πρόκληση, προετοιμασία της Γενικής Διεύθυνσης για νέους προσανατολισμούς για τη νέα περίοδο. Για την Ευρώπη 2020, αποτελέσματα και λοιπά. Αυτό θα σημαίνει αλλαγές και στα κράτη-μέλη και στην Κομισιόν τρίτη πρόκληση να βελτιωθεί η εφαρμογή στην φυστάμενη προγραμματική περίοδο και από πλευράς ουσίας και από πλευράς συμμόρφωσης γιατί έχουμε ακόμα κάποια ζητήματα όσον αφορά την ε, νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών. Ε, είμαστε καλύτεροι από τους παρελθόν, όπως βλέπετε από την τελευταία έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποια ζητήματα και το τρίτον, βεβαίω είναι και η ε, δυνατότητα απορρόφησης που πρέπει να βελτιωθεί. Τέταρτη πρόκληση, να βελτιωθεί η αξιολόγηση και η επικοινωνία και όλα αυτά με ε, λιγότερους εργαζόμενους. Οπότε είναι σαφές πως ε, με τέτοιες συνθήκες χρειάζεται αλλαγή του οργανισμού. Αλλαγή στο οργανόγραμμα, αλλά και αλλαγή στον τρόπο εργασίας. Οπότε υπήρχε πολύ υλικό που ήταν ήδη διαθέσιμο. Εμείς ως διοίκηση διαβουλευτήκαμε με τους ε, υπαλλήλους και αναπτύξαμε έτσι ένα σχέδιο το οποίο το λέμε αλλαγή ρέτζι. Και δεν είναι μόνο θέμα οργανογράμματος, είναι μια συνολική προσέγγιση θα έλεγα που συμπεριλαμβάνει τομείς όπως η αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, ενσωματώνει δηλαδή τις εσωτερικές μας διαδικασίες, αυξάνεται η παραγωγικότητα, αφορά τη διαχείριση της γνώσης, ε, εσωτερική επικοινωνία, περισσότερη προτεραιότητα στο βασικό μας έργο, καλύτερη διαχείριση του προσωπικού. Δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες, λίγα λόγια μόνο για την αναδιοργάνωση. Τα βασικά μπορούμε να τα συνοψίσουμε σε τρεις πτυχές. Πρώτα απ' όλα να γίνει πιο αποτελεσματικός ο οργανισμός και πιο μικρός. Δηλαδή είχαμε 10 διευθύνσεις, ε, τώρα έχουμε 8. Ήδη δηλαδή είμαστε πιο μικρός οργανισμός. Επίσης υπήρχαν ε, διάφοροι που περιφέρονταν ε, γύρω από τον Γενικό Διευθυντή, έχουν φύγει και αυτοί. Δεύτερον και σημαντικότερο, να ξεπεράσουμε αυτό το οποίο θα έλεγα είναι το οριζόντιο γεωγραφικό χάσμα. Με τα χρόνια είχε αναπτυχθεί ένα χάσμα μεταξύ αφενός των συναδέλφων που δούλευαν στην ανάπτυξη πολιτικής ε, και είχαν οριζόντια καθήκοντα συντονισμού και μετά υπήρχαν βεβαίως και τα γεωγραφικά γραφεία. Δεν κατηγορώ κανέναν γιατί και εγώ πριν από 8 χρόνια ήμουν διευθυντής οικονομικών και ήμουν μέρος ακριβώς αυτού του χάσματος. Αλλά εάν θέλουμε στο μέλλον να έχουμε έναν αναπροσανατολισμό της πολιτικής, τότε θα πρέπει το περιεχόμενο της πολιτικής να έρθει πιο κοντά στα προγράμματα. Γι' αυτό ακριβώς έγινε αυτή η αναδιοργάνωση. Τι κάναμε λοιπόν δημιουργήσαμε κέντρα αρμοδιοτήτων εντός των γεωγραφικών διευθύνσεων. Παραδείγματο χάρη, δύο κέντρα αρμοδιοτήτων για την Ευρώπη 2020. Ένα για την ε, έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη και ένα για την ε, ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή και βέβαια την ε, περιφερειακή διάσταση. Οπότε έχουμε και την Ευρώπη 2020 και την στενότερη συνεργασία μεταξύ της πολιτικής ε, πλευράς και της γεωγραφικής πτυχής. Και βεβαίως έχουμε και τρία άλλα κέντρα αρμοδιότητες. Ε, μία για τη διοικητική ικανότητα, μία για το ETC και αυτό το οποίο επίσης πρέπει να βελτιωθεί και εντός των κρατών μελών και της ε, Κομισιόν για μια επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα για να έχουμε μεγαλύτερη ε, παραγωγικότητα. Αυτό ήταν το δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο είναι πως βεβαίως δεν αλλάζονται, δεν αλλάζουν ε, όλα ταυτόχρονα και δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλουμε λοιπόν σταθερότητα μαζί με την αλλαγή. Σταθερότητα δηλαδή όσον αφορά τις σχέσεις με τα κράτη-μέλη και δεν αλλάξαν πολλά πράγματα ως προς αυτό, όσον αφορά δηλαδή τις ε, γεωγραφικές μονάδες. Βεβαίω, είναι πάρα πολύ νωρί να γίνει κάποια αξιολόγηση του νέου οργανογράμματος και Ναι, τέλος πάντων, ε, με τις ευκαιρίες να αναφερθώ και σε κάποια αποτελέσματα. Βεβαίως, όπως είπα, ε, που δεν σχετίζονται οπωσδήποτε με την αναδιοργάνωση. Όπως ξέρετε, στη γενική μας διεύθυνση πάντα ε, εργαζόμαστε σε τρεις χρονικές διαστάσεις στο παρελθόν, δηλαδή πρέπει να κλείσει η παλιά προγραμματική περίοδος, να εφαρμόσουμε τα εφιστάμενα προγράμματα και βέβαια να προετοιμάσουμε και το μέλλον. Δεν θα αναφερθώ στο μέλλον, γιατί εκεί έχουμε συνεχή διάλογο με τον Επίτροπο, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Πρόεδρο και τους συζητητές για τη φοβερή δουλειά που έχουν κάνει. Και νομίζω πως είναι πάρα πολύ θετικό το ότι ε, βλέπουμε πως εμείς είμαστε ο τομέας της ε, πολιτικής όπου έχει προχωρήσει περισσότερο η δουλειά στους κανονισμούς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λίγα λόγια τώρα για το ε, κλείσιμο. Όταν μιλάμε λοιπόν για τα προγράμματα 2000, 2006 έχουμε στείλει όλες τις ε, επιστολές ε, πλην 6. 277 ε, δηλαδή, πλην 377 πλην 6 επιστολών. 246 από αυτές αφορούν προγράμματα που έχουν κλείσει για τι υπόλοιπε, ε, βεβαίως ε, πρέπει να τα βρούμε με τα κράτη-μέλη. Οπότε βλέπουμε σαφώς πως υπάρχει φως ε, στο τέλος του τούνελ και αυτό δεν είναι μόνο διαδικαστικό ζήτημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία της πολιτικής έτσι ώστε να κλείσει η παλιά περίοδος. Είναι κάπως πιο πολύπλοκα τα πράγματα για τα ταμεία συνοχής γιατί βεβαίως εκεί πέρα πρέπει να κλείσουν έργο-έργο και αυτό το οποίο κάναμε είναι πως έχουμε μια ειδική ε, μονάδα που ασχολείται με το κλείσιμο των προγραμμάτων και βλέπουμε πως υπάρχει μια αύξηση της παραγωγικότητας. Για την τρέχουσα περίοδο ξέρετε πως λόγω της οικονομικής κρίσης έπρεπε να προσαρμόσουμε την πολιτική και τον προσανατολισμό της και αυτό σημαίνει βεβαίως και ένα προγραμματισμό για να αναφερθώ, για, ίσα ίσα για να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες που προέκυψαν με την κρίση, ειδικά όσον αφορά δηλαδή την ανεργία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε αν δει κανείς τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Από το 2009 έχουμε αναπρογραμματίσει 30 δισεκατομμύρια ευρώ, 25 εντός του ΕΤΠΑ και 5 στο ε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αναπρογραμματίζουμε ακόμα για την Ισπανία και Ελλάδα. Και αυτό το οποίο κάναμε είναι πως λάβαμε υπόψη και τις δυσκολίες των εθνικών προϋπολογισμών. Οπότε σε κάποιες περιπτώσεις μειώσαμε την εθνική συγχρηματοδότηση. Το θετικό λοιπόν είναι πως από τα στοιχεία ε, βλέπουμε ήδη ε, σημαντικά αποτελέσματα. Για να σας δώσω κάποια νούμερα για το 2011, γύρω στις 200.000 ε, θέσεις εργασίας αναφέρθηκαν από τα κράτη-μέλη ότι δημιουργήθηκαν από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής και άρα το σύνολο ανέρχεται σχεδόν στο διπλό σε 385.000. Ένα άλλο νούμερο 27.000 ε, νέες επιχειρήσεις που στηρίχθηκαν το 2011 και φέρνουν έτσι το σύνολο σε 53.000. Δείχνει αυτό νομίζω πως τα προγράμματα έχουν ήδη αντίκτυπο. Επίσης, τι είναι σημαντικό, τα διαθέσιμα κονδύλια να χρησιμοποιηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά και άρα το μήνυμα στα κράτη-μέλη και στις περιφερειές είναι απλό και διτό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επιλογής, ειδικά στους τομείς καινοτομίας, ΜΜΕ, σιδηροδρόμων, τηλεπικοινωνιών κτλ. Και βεβαίως να εφαρμοστούν και τα έργα τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει ή είναι, είναι σε εξέλιξη. Όπως ξέρετε, η εκτέλεση του προπολογισμού ποτέ δεν ήταν τόσο υψηλή από ό,τι στο τέλος ε, του έτου. Τελικά είχαμε ένα διορθωτικό προπολογισμό, αλλά δεν ήταν τόσο υψηλό όσο είχαμε ζητήσει. Αλλά ε, ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω και την Επιτροπή σας για την στήριξη για αυτά τα οποία υπέβαλε η Κομισιόν και ίσως χρειαστούμε και τη στήριξή σας ε, του χρόνου γιατί είναι ήδη σαφές πως ε, κάποιες ε, από τις αιτήσει πληρωμών που δεν θα καλύψουμε φέτος θα πληρώσουμε με πιστώση του επόμενο έτους. Οπότε τι κάνουμε. Εκεί όπου έχουμε ακόμα χρήματα πληρώνουμε πρώτα απ' όλα τις αιτήσει που ήρθαν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου για να σεβαστούμε τους δύο μήνες και η επόμενη προτεραιότητα είναι να πληρώσουμε τα προγράμματα που είχαμε μπλοκάρει και όπου ξεμπλοκάρουν τώρα και μετά έχουμε και τις χώρες ε, του προγράμματος ως επόμενη προτεραιότητα. Να αναφέρω τέλος πως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναφέρουν μέχρι το τέλος του έτους λεγόμενες εθνικές στρατηγικές αναφορές, το ότι έχουν επιτύχει και θα είναι σημαντική στιγμή για να αξιολογήσουμε και στο εθνικό και στο περιφερειακό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο της Ένωσης το πόσο καλά ε, έχουν επιτευχθεί αυτοί οι στόχοι σε περιφερειακό επίπεδο, ποιος ήταν ο αντίκτυπος της κρίσης, ποια ήταν η αντίδραση σε αυτήν, πώς τα προγράμματα συνεισέφεραν στην Ευρώπη 2020 και, πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη περίοδο, τι ε, διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Οπότε η Κομισιόν θα παρουσιάσει μια έκθεση το Μάρτιο και ευχαρίστως θα ξαναέρθω τότε στην Επιτροπή σας. Αυτά, κυρία Πρόεδρε, εν ολίγης, ε, για το τι γίνεται στο, στο μηχανοστάσιο της περιφερειακής πολιτικής Σας έδωσα κάποιες πληροφορίες για την εφαρμογή αλλά και τον εξυγχρονισμό της γενικής μας διεύθυνσης για να μπορέσει να προωθήσει ε, επιτόπου πολιτική για ανάπτυξη, για δουλειές στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όπως όλοι ξέρουμε ε, ζει την βαθύτερη κρίση της από το ξεκίνημά της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Διευθυντά Ολάμπερ Φανίστεροι. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ. Είναι παράδοση. Σε τακτά διαστήματα ο υπεύθυνο της Γενικής διάθεσης να έρχεται και να μας αναφέρει τα διάφορα σημαντικά θέματα για την πολιτική που κάνετε Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, μιλήσετε για επαναπροσω... επαναπροσανατολισμό. Είναι κάτι που έχει γίνει, γίνει, όλα έχουν λυθεί τα προβλήματα. Δεν υπάρχουν πλέον εντάσει. Αλλά κάτι χάθηκε. Τι είπατε. Υπάρχουν κάποια ε, προγράμματα, κάποια σχέδια που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Έγινε επαναπροσανατολισμός με απώλειες. Τι έγινε τέλος πάντων. Φερρυπίν. Πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου. Η συνοχή είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται σφαιρικά Πώς γίνεται η συνεργασία. Επίσης, είδα την εισήγηση που έγινε από την Ήτρα και αυτό το οποίο με εξέπληξε είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικές και Ανάπτυξης να μπορέσουν να επικοινωνήσουν σε επίπεδο κανονισμών και εκτέλεσής τους. Είναι πολύ διαφορετικά αυτά τα οποία γίνονται σε κάθε επίπεδο και για όλους ασχολούνται με το IT δεν μπορεί, όπως είπε ο Διευθυντής, να υπάρξει ένα διατάφτα, διότι είναι διαφορετικές οι ιδέες. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορείτε εσείς να συνεργαστείτε μεταξύ σας. Τι γίνεται σε επίπεδο εξωτερικής συνεργασίας. Και τι γίνεται με την αριστεία που θέλουμε να επιτύχουμε ακόμη σε επίπεδο των νέων κρατών και στα πλαίσια της πολιτικής 2020. Αυτά προς το παρόν. Ο Γιάνν Όλμπριχτ. Σα ευχαριστούμε, κύριε Γενική Διευθυντά, που ήρθατε και αν είναι δυνατόν να μας στείλετε το νέο σας οργανόγραμμα, διότι μας περιγράψατε κάποια πράγματα και κάποια άτομα, αλλά καλύτερα να το έχουμε και γραπτός. Εάν ήδη έχει εγκριθεί και το έχετε γραπτός. Έχω για τα αστικά θέματα κάποιες ερωτήσεις. Διότι ασχολείστε από την 1η Δεκεμβρίου και με θέματα, όπως λέγεται, περιφερειακά και αστικά. Τι σημαίνει αυτό εκτός από το όνομα στην πράξη. Υπάρχει μονάδα που ασχολείται με αστικά θέματα. Επίσης, τα πλαίσια της Προεδρίας Κυπριακής και της ε, ε, Ιρλανδικής Προεδρίας μιλάτε για urban platform, για ε, βήμα αστικό. Τι σημαίνει αυτό. Τι γίνεται επίσης σε επίπεδο ε, ένας Δημάρχων, τι γίνεται επίσης με τις ευφυείς πόλεις όπως λέγονται στα θέματα ενεργειακά. Ξέρω ότι ένα από τα κέντρα αυτά έχει σχέση με την ε, ενέργεια και μέχρι τώρα όλα αυτά ήταν θέμα, μέχρι τώρα με αυτά τα θέματα ασχολείται η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Επίσης, θα αλλάξετε και το ακρονίμιο. Τι σημαίνουν όλες αυτές οι αλλαγές που μας αναγγείλατε στην πράξη. Ο Ιωαχήμ Τσέλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Γενικό Διευθυντή. Θέλω να υπογραμμίσω αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Λάμπερτς. Χρειάζεται μια διοργανική συνεργασία και εντός της Γενικής Διεύθυνσης αλλά και μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων. Βλέπουμε πως εγκρίνονται και εντός του Κοινοβουλίου από διάφορες επιτροπές, διάφορες εκθέσεις και όταν λένε πού θα βρουν τα λεφτά λένε «Α, στα διαρθρωτικά ταμεία». Βεβαίω δεν πάει έτσι. πρέπει ήδη εντός της Κομισιόν να είναι ξεκάθαροι οι κανόνες του παιχνιδιού και τα υπόλοιπα μέλη και οι υπάλληλοι της Κομισιόν να ξεκαθαρίσουν ε, στις υπόλοιπες επιτροπές ε, πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα λεφτά και πού όχι. Αναφερθήκατε στο ότι έχουν ε, τυπωθεί επιστολές ήδη, έχουν αποσταλεί επιστολές ήδη ε, για αυτή την περίοδο. Μα εργαζόμαστε ήδη για την περίοδο 14 έως 2020 και σήμερα ε, βλέπουμε πως η κατάσταση Δεκέμβριος ε, του 2012 είναι κάπως ανησυχητική. Συζητήσαμε πριν και με την Κυπριακή Προεδρία και εκεί πέρα τόνισα πόσο σημαντική είναι η διαρθρωτική πολιτική ως μια πολιτική της εσωτερικής συνοχής και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Τα νούμερα αυτά όμως σχηματίζουν μια εικόνα σύμφωνα με την οποία τα οικονομικά ισχυρά κράτη διαχειρίζονται καλά τα κονδύλια τους και είναι τα στενέστερα κράτη που έχουν ακριβώς ε, μεγάλα ελλείμματα σε αυτό το τομέα. Και ε, πρέπει να ξαναδούμε το όλο ζήτημα της πολιτικής συνοχής, γιατί υπάρχουν κράτη-μέλη που αμφισβητούν το νόημα τη πολιτικής συνοχής και θέλουν άλλε μεθόδους. Διαβάζω εδώ πέρα πως κάποια κράτη έχουν απορρόφηση 20 με 30% των διαθέσιμων κονδυλίων. Και αναρωτιέμαι τι θα γίνει στο μέλλον. Είχαμε και τώρα τη συζήτηση ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός δεν μπορεί να εκπληρώσει τις ε, πληρωμές του γιατί ε, τώρα έχουμε περισσότερες πληρωμές ε, από το ετήσιο πλαφόν. Οπότε θα πρέπει ίσως να μοιράζονται τα κονδύλια σε ολόκληρη την πραγματική περίοδο, αλλά βέβαια υπάρχει μετά το πρόβλημα που αναφέρθηκε με την ε, Προεδρία του Συμβουλίου. Δηλαδή, εάν η συζήτηση για τον κανονισμό και τη χρηματοδότηση του Πουδουπού πάει πιο πολύ στο μέλλον, τότε βεβαίως ε, καθυστερούμε και τη διαδικασία της εφαρμογής και το πρόβλημα θα είναι στις ε, περιφέρειες που δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν αυτή τη στιγμή ανέφερα πως ε, σε πολλές περιφέρειες έχουν επιτροπές ε, παρακολούθησης αλλά έχουν αναστείλει το έργο τους γιατί δεν ξέρουν πώς θα διαμορφωθεί τελικά ο κανονισμός. Πώς μπορεί λοιπόν εδώ πέρα να παρέμβει η Κομισιόν για να στηρίξει ειδικά εκείνα τα κράτη-μέλη που μέχρι στιγμής είναι πολύ πίσω από τα υπόλοιπα όσον αφορά την ε, την απορρόφηση και τη χρήση των, των κονδυλίων. Κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ ε, για την παρουσίαση που μας κάνατε. Εγώ θα σας κάνω μια γενικότερη ερώτηση αν μου επιτρέπετε. Ε, μιλήσατε και εσείς για ανάπτυξη και είναι προφανές σε όλους μας ότι η πολιτική συνοχής, αν την έχω καταλάβει καλά, αποσκοπεί στο να ε, υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή οι ανισορροπίες να εξαλειφθούν με την πάροδο του χρόνου και να έχουμε μια ε, σχεδόν ανάπτυξη στο ίδιο επίπεδο. Λίγο Αυτό σημαίνει και cohesion. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Με αυτά τα δεδομένα και με, με δεδομένο ότι υποτίθεται ότι προωθείται μια πολιτική συνοχή. Εσείς πώς εξηγείτε το γεγονός ότι παραδείγματο χάρη οι ανισότητες στο εσωτερικό της Ελλάδας για την οποία είμαι σε θέση να μιλήσω έχουν αυξηθεί παρά την εφαρμογή της cohesion policy. Αυτά δείχνουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερη ερώτηση. Πώς εξηγείτε εσείς ε, μια διαπίστωση που είχε γίνει σε μια ε, θεώρηση του Ταμείου Συνοχής όσον αφορά τους δρόμους και όσον αφορά έργα για την προστασία του περιβάλλοντος, όπου για τους μεν δρόμους υπόθηκε ότι μόνο οι δρόμοι δεν οδήγησαν σε ανάπτυξη, εκεί που αναπτύχθηκαν οι δρόμοι, και τα δε χρήματα για το περιβάλλον, τα έργα για το περιβάλλον, γίνανε κυρίως για να προσαρμοστεί η νομοθεσία των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών στο κοινοτικό και εκτιμένο. Κλείνω με το εξής ερώτημα. Ε, μιλήσατε και εσείς, αλλά όχι μόνο εσείς, ξέρω ότι είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά. Ευρώπη 2020. Υπάρχουν ε, προγράμματα προσωμείωσης στη διεύθυνσή σας που να δείχνουν ότι πράγματι, εάν η Ελλάδα εφαρμόσει στο ακέραιο του στόχου της Ευρώπης 2020 το 20 θα έχει αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 10, 5, 3, 1, πόσο της εκατό. Θα αυξηθεί πιο γρήγορα στην Ελλάδα από ό,τι στη Γερμανία λέμε για να φτάσει στο ίδιο επίπεδο με Ευρώπη 2020. Όχι με άλλα. Με Ευρώπη 2020. Διότι εγώ ισχυρίζομαι ότι με Ευρώπη 2020 θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η απόσταση και είναι πάρα πολύ απλό, δεν θέλει καμία θεωρία. Ευρώπη 2020 προϋποθέτει χρησιμοποίηση και ανάπτυξη συγκεκριμένων τεχνολογιών που οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες δεν τις έχουν και ούτε πρόκειται να μπορέσουν ποτέ να τις αναπτύξουν. Τελειώνω με το, με το ερώτημα το εξή. Υπάρχουν προγράμματα προσωμείωσης στη διεύθυνσή σας που να μπορούν επιστημονικά να τεκμηριώσουν αυτές τις επιλογές που κάνετε. Ναι ή όχι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Director, the floor is yours. Έχετε το λόγο κύριε Δευθυντά. Well, thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Ελπίζω ότι τα σημείωσα όλα. Κύριε Βανίστελ Ροϊ, Ζητήσατε να έχουμε απώλειες με τη νέα μας οργάνωση. Χάσαμε δύο θέσεις διευθυντών. Είχαμε δέκα διευθυντές και τώρα έχουμε οκτώ. Αλλά αλλά δεν χάσαμε ε, καθήκοντα το πρέπει να φέρουμε σε πέρας. Και μεθαύριο πρέπει να σας πω θα πάω στην Κίνα αντικαθιστώντας τον Επίτροπο. Άρα από αυτά τα οποία είχαν ανατεθεί στη μας δεν χάσαμε τίποτε. Αυτό το οποίο θα κάνουμε, και αυτό νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον είναι ότι δεν κάνουμε τα πάντα μόνοι μας. Θα χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο πραγματονόμους, οποίους θα αναθέτουμε κάποιες αποστολές. Διότι, όπως σας είπα, θα χάσουμε προσωπικό. Κάθε χρόνο θα χάνουμε κάποια άτομα. Αλλά πρέπει να την αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, όντας και πιο παραγωγική Άρα θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να συνεργαστούμε και με άλλες γενικές διευθύνσεις στο τομέα του οικονομικού ελέγχου, εσωτερικού οικονομικού ελέγχου. Θα παίξουμε περισσότερο με τις συνέργειες από ό,τι σήμερα, για είμαστε πιο αποδοτικοί. Θα αναθέσουμε και σε εξωτερικούς συνεργάτες δηλαδή κάποια πράγματα από αυτά που πρέπει να κάνουμε στην γάμα δέλτα μας. Σωστός λοιπόν και έπρεπε να το είχα αναφέρει το όνομα της Γενικής μας Διεύθυνσης άλλαξε. Είμαστε η περιφερειακή και αστική πολιτική. Ρέτζι όμως είναι η... το ακρονίμι. δεν έχει αλλάξει. Και μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας και να δείτε το νέο μας οργανόγραμμα. Και αν θέλετε, μπορούμε να σας στείλουμε και να τυπώσουμε τα αντίγραφα. Ούτως ή όλα αυτά δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας. Είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία και μπορείτε να δείτε ότι τα βασικά λειτουργίε και καθήκοντα που μας είχαν ανατεθεί καλύπτονται. Επίση, η συνεργασία μεταξύ των διαφορών γάμα είναι κάτι που ερωτήσατε. σε σχέση με την έρευνα και την περιφερειακή πολιτική. Μία από τις κύριες διαφορές είναι ότι η γάμα δέλτα μας συνεργάζεται πολύ περισσότερο από το παρελθόν με τις άλλες γάμα δέλτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δείτε και στην Παπασκευή της επόμενης περίοδου. Έχουμε, ε, περίοδο, έχουμε διάφορες κοινέ ομάδες, για θέματα περιφερειακής ε, συμπερίληψης, για θέματα ε, εφιών πολιτικών που θα εφαρμόσουμε. Η JRC έχει και ένα ε, βήμα στην Σεβίλη για να υποστηριχτούν αυτές οι νέες στρατηγικές οι δύο λοιπόν γάμα δέλτα μας συνεργάζονται και προσπαθήσαμε να βρούμε και τρόπο για να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε τις δύο πολιτικές. Yeah. So, ώστε να μπορέσουμε να βαθίσουμε προς την πολιτική της αριστείας στα πλαίσια της συνεργασίας μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται προς τις δύο κατευθύνσεις. Και πριν και μετά. Διότι στην Ευρώπη αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να μπορέσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας να τα εφαρμόσουμε στην καινοτομία και στην ε, πράξη. Η πολιτική μας, λοιπόν, πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει με την καινοτομία, την υποστήριξη των ΜΜΕ και τα λοιπά. Υπάρχει, λοιπόν, πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των δύο τομέων αυτών. Και αυτό δεν αφορά μόνο την έρευνα, αλλά και τις μεταφορές, την ενέργεια και άλλες. Ανέφερε ο κ. Σόλμπρικ την διάσταση αυτό το αστικό που είπαμε, γιατί άλλαξε το όνομα. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, για να είναι αναγνωρίσιμη η σημασία του αστικού σκέλους, του αστικού στοιχείου. Γι' αυτό προσθέθηκε αυτό στην τίτλο της ΓΔ και δεύτερον, διότι στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ εμείς έχουμε σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε στα πλαίσια του συντονισμού των διαφόρων πολιτικών. Τον προηγούμενο μήνα προείδρευσα μία συνεδρίαση ε, μεταξύ όλων των υπηρεσιών και γενικών διευθύνσεων συγγνώμη, με τις οποίες συνεργαζόμαστε και είπαν ότι πρέπει να είμαστε πιο συντονισμένοι. Διότι θα πρέπει να έχουμε πολύ καλή διασύνδεση και συντονισμό και τον βγαίνουμε και εκτός να ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα. Πρόκειται για σημείο όντως και βεβαίως θα πρέπει να εργαστούμε για μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ όλων ημών. Και του χρόνου θα δούμε πώς μεταξύ μας όλοι θα μπορέσουμε να εντάξουμε και αυτή τη διάσταση, την αστική αν θέλετε, την αστική πολιτική που θέλουμε να κάνουμε σε όλες τις πολιτικές μας. Όλα αυτά σε ένα πολύ θετικό πνεύμα συνεργασίας. Κύριε Τσέλερ, αναφερθήκατε στο πρόβλημα της απορρόφησης στα ασθενέστερα κράτη-μέλη. Είναι μια ανησυχία δική μας επίσης. Και δικαίως νομίζω έχουμε πει πως υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη όπου έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα απορρόφησης. Το ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα ήταν άλλος ένας λόγος ε, για το ότι ακριβώς φτιάξαμε και ένα κέντρο αρμοδιότητας για διοικητική ικανότητα και το κάνουμε αυτό ήδη στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, δηλαδή ε, με την ε, Παγκόσμια Τράπεζα, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης συνεργαζόμαστε για να εξοπλίσουμε αυτά τα κράτη-μέλη με ε, διοικητική ικανότητα. Επίσης ε, δίνουμε κάποια βοήθεια στα κράτη-μέλη για την προετοιμασία ε, των επόμενων περίοδων. Όπως ξέρετε, όλες οι υπηρεσίες της Κομισιόν, άρα και αυτές οι οποίες ασχολούνται και για το πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά και εκεί πέρα όπου καταρτίζονται τα position papers, παρουσιάζουμε ακριβώς το τι εμείς θεωρούμε πως είναι οι σημαντικότερες προτεραιότητες για τα ταμεία αυτά στο μέλλον και σε αυτά τα έγγραφα θέσεων ε, φύγεται το ζήτημα της ε, διοικητικής ικανότητας. Ε, είναι ακόμα ένα ζήτημα πάνω στο οποίο εργαζόμαστε. Κύριε Αγκουράκη, αναφερθήκατε σε προβλήματα μη αποτελεσμάτων. Ε, είναι κάπως μονομερές αυτό το οποίο λέτε. Υπάρχουν προβλήματα εδώ και εκεί, αλλά αν δείτε τη γενική αξιολόγηση, είναι σαφές πως υπάρχουν αυξήσεις στο ΑΕΠ ε, που φαίνονται μέσω της οικονομικής ανάλυσης. Έχω ένα στοιχείο πρόχειρο, νομίζω για τα νέα κράτη-μέλη είναι γύρω στο 1,2% του ΑΕΠ σε σύγκριση έτσι με κάποιο σταθερό σημείο αναφοράς. Γιατί αυτό το οποίο βλέπετε στην πραγματικότητα βεβαίω είναι πάντα, οφείλεται πάντα σε πολλούς παράγοντες. Ε, αν απομονωθεί μόνο η πολιτική συνοχή, βλέπετε θετικά αποτελέσματα. Ε, δύο άλλα σημεία αναφέρατε. Έτσι επικριτικά. Το ένα αφορούσε τις περιβαλλοντικές επενδύσεις, ότι δηλαδή αφορούν το να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη για να επιτύχουν τις υψηλότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ε, δεν είναι σκάνδαλο αυτό. Είναι θετικό το ότι η πολιτική συνοχής βοηθάει τα κράτη-μέλη να επιτύχουν υψηλότερες προδιαγραφές. Αν δεν το κάναμε αυτό, τι αποτέλεσμα θα είχαμε. Τα κράτη-μέλη δεν θα δέχονταν υψηλότερες προδιαγραφές και αυτό θα ήταν εις βάρος ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν νομίζω πως πρέπει να είμαστε πολύ επικριτικοί στο να βοηθάμε τα, τα κράτη-μέλη ε, να επιτύχουν τις προδιαγραφές αυτές. Για την καινοτομία. Η έννοια της καινοτομίας δεν είναι μόνο υψηλή τεχνολογία. Υπάρχει πολύ καινοτομία στις διαδικασίες, στα προϊόντα, σε οποιοδήποτε επίπεδο μπορεί να υπάρχει καινοτομία στον τουρισμό, χωρίς υψηλή τεχνολογία. Πρέπει λοιπόν να δούμε ευρύτερα την καινοτομία. Εμείς αυτό προωθούμε. Η καινοτομία είναι το να προσαρμόζεται κανείς αλλαγές στην αγορά, να έχει νέες ιδέες, κοινωνική καινοτομία, παραδείγματο χάρη. Ναι. Είναι λοιπόν κάτι το, το ευρύτερο από την υψηλή τεχνολογία. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να απάντησα λίγο πολύ στις ερωτήσεις των βουλευτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Απευθύνομαι στους αριστές. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσω τη μέθοδο DONT. Ελπίζω να μην σας ενοχλεί αυτό ιδιαίτερα. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε γιατί δεν έχουμε άλλες παρατηρήσεις. Ελπίζουμε να ξαναδούμε το Φεβρουάριο-Μάρτιο, μας είπατε, όταν θα είναι έτοιμη έκθεση, το Μάρτιο. Πολύ ωραία. Εκτός ο, μικροφώνου κ. Μποστινάρου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, τα όσα είπατε για την Κίνα εκ το ταξίδι σας στην Κίνα με έκανα να κάνω την ερώτηση αυτή. Η Γενική Διεύθυνση Ρέιτζιο είναι μέρος της εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Αν ισχύει κάτι τέτοιο θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί εδώ και πάρα πολλούς μήνες είχα δώσει πραγματικό αγώνα εγώ με τον κύριο Βανιστερό για κάτι τέτοιο. Δεύτερη ερώτηση. Η Γενική σας Διεύθυνση μπορεί να βοηθήσει πλέον την Ρουμανία για την ε, οικοδόμηση θεσμών στη χώρα μέσω της νέας σας οργάνωσης προκειμένου να υπάρχει μια καλύτερη χρησιμοποίηση των κοινοτικών πόρων και μπορείτε να βοηθήσετε τη ρουμανική κυβέρνηση προκειμένου να εφαρμοστεί η περιφερειακή, νέα περιφερειακή πολιτική το 2013. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να συναφερθώ πάλι στην Κίνα. Προφανώς ένα από τα βασικά ζητήματα που θα συζητήσουμε στην Κίνα είναι η σχέση ανάμεσα στις πόλεις, την Ήπεθρο, πώς μπορούμε να διασυνδέσουμε τους δύο αυτούς τομείς. Ξέρετε ότι ε, έχουμε και ένα πρόγραμμα ανταλλαγών. Πολλές φορές ε, Κινέζοι εκπρόσωποι έρχονται και στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι σε κάτι τέτοιο πρέπει να αναφερθήκατε. Για να είμαι όμως ειλικρινής, ανησυχώ περισσότερο για τη Ρουμανία. Κύριε, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη που διακόπτω. Μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, να πάρω το λόγο, λέει ο κύριος Βανίστερο. Ναι, έχει ολοκληρώσει ο Βίκτορ. Εκτός μικροφώνου. Λοιπόν, να σας ακούσουμε τον Λάμπερτ. Είπατε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τα προγράμματα. Εμείς όμως συμμετείχαμε στα προγράμματα αυτά και βλέπουμε ότι η Γενική σας Διεύθυνση έχει εγκαταλείψει κάποια προγράμματα. Τα έδωσε προς την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Το σημαντικό είναι ότι η κυρία Χούμπνερ ξεκίνησε τα προγράμματα αυτά. Αυτή ξεκίνησε αυτόν τον διάλογο και γίνανε κάποιες καταπληκτικές αναλύσεις για την ε, πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την πολιτική που ακολουθεί η Κίνα. Ο πρώην συνάδελφός σας ε, στην περιοχή του ε, Σετσουάν στην Κίνα προσπαθεί πραγματικά να βοηθήσει τους εκεί θύνοντες με μια πολιτική συνοχής. Πηγαίνει επίσης στην Κίνα και ο Μπαρόσο και μιλάει όμως μόνο για την πολιτική περιβάλλοντος. Μ' αρέσει αυτά τα οποία λέει, αλλά μ' αρέσουν αυτά τα οποία κάνετε εσείς περισσότερο. Είναι σημαντικό λοιπόν όμως να αναλάβετε δράση και να αναλάβετε τις ευθύνες σας, γιατί έχω την εντύπωση ότι σιγά σιγά εγκαταλείπεται αυτή την πολιτική. Στο Intergroup για την αστική πολιτική στις, στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά δυστυχώς εσείς δεν έχετε ανάλογη δράση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας προτιμάτε σε σχέση με άλλους, λέει ο κύριος Δεφά. Ξέρω βέβαια ότι η προτίμηση αυτή δεν θα πρέπει να θεωρώ δεδομένη. Σας εξασφαλίζω, ε, σας λέω πάντως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα συντονιστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμείς για τα ζητήματα αυτά. Αληθεύει όμως και αυτό το οποίο μόλις τώρα είπα, ότι η Ρουμανία είναι πιο σημαντική για μένα από ότι είναι η Κίνα. Ωστόσο βέβαια θα πάω στην Κίνα. Επανέρχομαι όμως τώρα στα όσα έλεγα για τη Ρουμανία. Είμαστε σε πολύ στενή επαφή με τους συναδέλφους από τη Ρουμανία. Ξέρετε ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου εύκολη. Και αυτό γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα στη Ρουμανία όσον αφορά το ζήτημα της συμμόρφωσης και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την διοικητική ικανότητα της χώρας. Συνεπώς, ήδη αύριο θα μιλήσω με τον Αντιπρόεδρο της Παγκοσμίου Τράπεζας και ένα από τα ζητήματα που θα συζητήσουμε είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα την ρουμανική διοίκηση να δημιουργήσει τις απαραίτητες ικανότητες προκειμένου να απορροφήσει τα κοινοτικά κονδύλια. Αυτό ξέρετε ότι πάει παραπέρα από την απλή διαχείριση των κονδυλίων. Ουσιαστικά αναφερόμαστε εδώ πέρα στην αναδιάρθρωση ολόκληρων πολιτικών, όπως η πολιτική για το είδωρ ή η πολιτική για τις μεταφορές. Πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη πολιτική διάρθρωση, η οποία θα είναι σε θέση να απορροφήσει τα κοινωτικά κονδύλια στη συνέχεια. Αυτή είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες και αντικατοπτρίζεται αυτό στη νέα αυτή μονάδα που έχουμε, που ασχολείται με το ζήτημα της διοικητικής ικανότητας θεωρώντα το μία από τι βασικέ αρμοδιότητε πρέπει και εμεί να προωθήσουμε από τη δική μα Γενική Διεύθυνση. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Αν δεν υπάρχουν άλλε ερωτήσει παρατηρήσει, να ευχαριστήσουμε τον Γενικό Διευθυντή και ελπίζουμε να σα ξαναδούμε εδώ σύντομα. Στο ενδιάμεσο διάστημα, ο Νίκολα ε, Μάρτιν θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις και ξέρετε ότι σας υποβάλλει αναφορές, επομένως εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τι συζητάμε και εμείς εδώ και όπως βλέπουμε και στην τεχνική συνεργασία που θα έχουμε και τον επόμενο μήνα. Γιατί ξέρετε ότι χρειαζόμαστε αυτή την τεχνική υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Επομένω, ε, στηριζόμαστε όχι μόνο στην ενεργό συμμετοχή σα εδώ, αλλά και στο να μα βοηθάτε μέσω τη τεχνική σα εμπειρογνωμοσύνη να καταλήγουμε και εμεί σε κάποιε συμφωνίε και συμβασμού. Ο κύριο Ντεφά. Το μόνο το οποίο θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή είναι πως η διοίκηση, ο Νικολάς Μάρτιν και εγώ θα κάνουμε όλα όσα χρειάζεστε για τις επιτυχείς διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό. Νομίζω πως ε, πάμε προς σωστή κατεύθυνση. Και δεν είναι μόνο ζήτημα παρουσίας. Ξέρετε πως, ε, πόσο εμπλέκεται ο Νικόλας στην τεχνική πτυχή και παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεστε προς συμφέρον όλων μας και της ε, πολιτικής της περιφερειακής. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, θα συνεδριάσουν οι συντονιστές. Όσοι λοιπόν δεν θα μείνουν σε αυτή τη συνεδρίαση, παρακαλώ να φύγουν από την αίθουσα. Ε, Και όσοι δεν είναι εδώ, αν μπορεί κάποιος να τους ζητήσει να έρθουν το στομό το δυνατό.